So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίζω όσους ήταν και χθε το βράδυ εδώ και όλους τους υπόλοιπους εκπροσώπους της Κομισιόν. Πρώτα πρώτα να ρωτήσω εάν υπάρχουν παρατηρήσεις για την ημερήσια διάταξη. Θέλετε κάτι να αλλάξει. Όχι. Οπότε εγκρίνεται. Σήμερα έχουμε ένα πιο χαλαρό πρόγραμμα. Μετά θα αλλάξει με την ε, απαλλαγή όταν θα πηγαίνουμε προς την ψηφοφορία. Λοιπόν, για τις ανακοινώσεις ε, έχουν, έχουμε όλες τις γλώσσες που έχουν ζητηθεί. Μετά έχουμε τις συστάσεις των ε, συντονιστών της 23ης Ιανουαρίου και 21ης που 23 σας μοιράστηκαν. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Όχι. Οπότε συνεχίζουμε. Μετά έχουμε την αποστολή στην ε, τσεχική δημοκρατία να σας ρωτήσω εάν ε, θέλετε να γίνει κάτι, κάποια αλλαγή. Η Κομισιόν έκανε κάποιες ε, παρατηρήσεις. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις της Κομισιόν για το πού πρέπει να πάμε. Ή από τη μεριά του Όλαφ, αν υπάρχει κάποια πρόταση ή επιθυμία. Βεβαίως ε, δεν είμαστε εμείς ε, ελεγκτές, είμαστε πολιτικοί και ως πολιτικοί πηγαίνουμε στην αποστολή, οπότε δεν έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα να κάνουμε μια πραγματική αξιολόγηση, οπότε πρόκειται για μια πολιτική ε, αποστολή, να κάνουμε ερωτήσεις για τα συστήματα και δεν θα μπούμε σε λάθος ρόλο. Λοιπόν, υπάρχουν... Υπάρχει κάτι το οποίο θα θέλατε να δούμε, απευθύνομαι στην ε, Κομισιόν ή στον ε, Όλαφ, ε, η κυρία Μπόρχμαν νομίζω θα μπορούσε να μας απαντήσει. Das That is much better, I think. Thank you, Chair. Sorry for waking you up like... Ναι, πολύ καλύτερα. Συγγνώμη που έκανα αυτή τη φασαρία και σας ξύπνησα. Να σας ευχαριστήσω για την διευκρίνηση ότι πράγματι είναι μια πολιτική αποστολή, μια διερευνητική επιστολή την οποία διοργανώνεται. Προφανώς όταν οι ελεγκτές αξιολογούν τη συμμόρφωση, αυτό γίνεται βεβαίως στο πλαίσιο των εξελισσόμενων ελέγχων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή γίνονται στην Τσεχία. Όσον αφορά προτάσεις για το τι θα κάνετε, από ελεγκτική πλευρά θα έλεγα να μην πάτε εκεί που έχουμε κάνει ήδη ελέγχου. Γιατί ακριβώ βρίσκονται σε εξέλιξη ορισμένοι έλεγχοι. Οπότε αυτό θα είχα να σα πω εγώ σαν σύσταση. Αν θέλετε, μην πάτε σε αυτά τα έργα που έχουν καλυφθεί ήδη από δικούς μας ελέγχους. Κατά τα άλλα, από το σχέδιο προγράμματος που έχω δει, βλέπω ότι έχετε σκοπό να συναντηθείτε με διάφορες μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Βλέπω ότι θα έχετε και συναντήσεις με εθνικές αρχές και με οργανισμούς ε, πληρωμών με τους οποίους ασχολούμαι εγώ στη δουλειά μου. Αυτό βεβαίως είναι δική σας ε, επιλογή, το με ποιον θα συναντηθείτε και σε παλαιότερες ε, αποστολές σας έχετε συναντηθεί με οργανισμούς πληρωμών που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των, αγροτικών, των γεωργικών κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Από αυτή την άποψη δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πάτε και να τους συναντήσετε. Απλά για να, ε, για να είναι ξεκάθαρος, λέω εγώ, ο, ο σκοπός αυτής της αποστολής. Όσον αφορά προτάσεις, δηλαδή συγκεκριμένες για το με ποιον θα ήταν καλό να μιλήσετε, να συναντήσετε. Εσείς είστε βεβαίως ε, οι πρώτοι αρμόδιοι για να το αποφασίσετε. Θέλω να πω κάτι πολύ ε, προσεκτικά να σας πω το εξής. Αυτό που λέτε δεν γίνεται. Γιατί πρώτον δεν ξέρουμε ποιους έχετε ελέγξει Οπότε δεν μπορούμε και να αποφύγουμε άτομα τα οποία έχετε υποβάλει εσείς σε έλεγχο. Επίσης, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό, προφανώς και για την Επιτροπή μας είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο το ενδιαφέρον να πάμε ακριβώς εκεί. Όχι να πάμε εκεί που δεν υπάρχουν προβλήματα. Αντιθέτω, ε, μας καλούν οι πολίτες ή περιμένουν από εμά οι πολίτες να πάμε εκεί όπου υπάρχουν προβλήματα. Οπότε θα μας απασχολήσουν και αυτά τα προβληματικά θέματα, αν θέλετε. Ανεξάρτητα τελείως από τους δικούς σας ε, ελέγχους. το έχουμε κάνει στο παρελθόν και στη Σλοβακία έτσι. Δεν καθορίζουμε την ατζέντα μας ε, με βάση το πού γίνονται έλεγχοι, αλλά το πού και, που, και με ποιους πρέπει να συναντηθούμε στο πλαίσιο ε, μιας τέτοιας ε, επίσκεψης αποστολής. Θα ήταν και περίεργο να πηγαίναμε μόνο εκεί όπου δεν υπάρχουν προβλήματα. Θα ήταν μια τουλάχιστον περίεργη στάση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εμείς έτσι τις διοργανώνουμε πάντοτε αυτές τις ερευνητικέ ε, αποστολές και έτσι θα το κάνουμε και αυτή τη φορά. Ωραία, Ήλζε Βαντενάλμπετ που είναι τμήματάρχης για τους ε, λογιστικούς ελέγχους κομισιών. Ευχαριστώ. Από την DG Regio. Είμαι υπεύθυνη για τους ελέγχους για τη σύγκρουση συμφερόντων στην Τσεχία. Θέλω να θέσω, να ε, να σας ζητήσω δύο πράγματα. Πρώτον, να ξεκαθαρίσετε τον τίτλο της αποστολής, γιατί για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά την αξιολόγηση του, των, της αποτελεσματικότητάς τους για ε, την... Ε, για την εξασφάλιση το, της ορθής χρήσης των κονδυλίων. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε κάνει ήδη. Να ξεκαθαρίσετε δηλαδή ότι δεν κάνετε έλεγχο εσεί, αλλά ότι είναι μια ερευνητική αποστολή. Δεύτερον, θα θέλαμε... προέδρο. ναι, το έχουμε ξεκαθαρίσει ήδη πέντε φορέ. Συνεχίζει η ομιλήτρια. Θέλουμε να σα βοηθήσουμε στη συνάντησή σας με την ελεγκτική αρχή, γιατί βλέπω ότι και στο πρόγραμμά σας προβλέπετε κάτι τέτοιο και οι συνάδελφοί μας είναι βεβαίως στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια χρειάζεστε κατά τη διοργάνωση της αποστολής αυτή. Σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος, ε, να επιδεικνύετε σεβασμό στο Κοινοβούλιο, γιατί είναι και δική μας αρμοδιότητα. Έχουμε κάνει το ίδιο και στη Σλοβακία και σε άλλες χώρες και στην Ελλάδα. Έχω συμμετάσχει σε πολλές αποστολές. Θα ήταν ε, τουλάχιστον περίεργο να μην αγγίζει η Επιτροπή μας τα προβληματικά θέματα. Οπότε νομίζω ότι και μια επιστροφή στην κανονικότητα ε, δεν θα ήταν κακή. Αυτά κάνουμε συνήθως. Οι ερευνητικέ αποστολές που κάνει το Κοινοβούλιο είναι κάτι εντελώς συνηθισμένο και φυσιολογικό. Αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ και για τη βοήθεια που μας ε, προσφέρετε. DG Empl, Mark Sheffield, εκτελεστικός διευθυντής. Δεν ακούω κάτι, οπότε μάλλον δεν είναι μαζί μας. Από τον Όλαφ έχουμε μαζί μας τον κύριο Ερνέστο Μπιάνκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Είδα το πρόγραμμα που προβλέπετε. Μια χαρά είναι. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε να σας βοηθήσουμε, ευχαρίστω και θα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ε, τα θέματα τα οποία θα διαπιστώσετε στην αποστολή αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και που ασχοληθήκατε σε βάθο με τα ζητήματα και τα πορίσματά μας από την αποστολή, από την αποστολή στην Σλοβακία όπου νομίζω ότι και η δική μας Επιτροπή συνέβαλε στην διαμόρφωση, διαμόρφωση μιας νέας οπτικής, αν θέλετε, για τα πράγματα. Δεν ήταν πάντοτε ευχάριστη αυτή η δουλειά της Κοντ, αλλά και όλα αυτά τα ίδια δυσάρεστα καθήκοντα εκτελεί από διαφορετικό πρίσμα βεβαίως και από διαφορετική θέση από ότι μια κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά σας ευχαριστούμε και πάλι για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Συνάδελφοι, υπάρχουν ε, ερωτήσεις ή άλλες συστάσεις όσον αφορά την διοργάνωση αυτής της αποστολής. Ωραία. Άρα θα προχωρήσουμε έτσι όπως ε, προκύπτει από τη σύσταση των συντονιστών. Δεν βλέπω να υπάρχουν αλλαγές, ούτε ως προς το χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί. Η κυρία Στουργάριου. Ναι, συζητούσαμε μήπως το συζητήσουμε και σε επίπεδο συντονιστών, το ξέρω ότι έχει συζητηθεί στη διάσκεψη του Πρόεδρου. να υπάρχει ένα ψήφισμα μετά την ε, ερευνητική αυτή, διερευνητική αυτή αποστολή, στο οποίο θα συμπεριληφθούν όλα τα πορίσματα που θα προκύψουν από την αποστολή. Ναι, θα το συζητήσουμε, λέει η Πρόεδρος, με τους συντονιστές. Έχει ξανακαταβληθεί αυτή η, η, πρόταση, δεν είναι πρώτη φορά. Πρέπει όμως βεβαίως να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί πρέπει να αποφασιστεί κάτι τέτοιο στη διάσκεψη των ε, Προέδρων σχετικά γρήγορα για το πότε θα μπορούσε να γίνει αυτό το ψήφισμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη συζητήσει. Οπότε και εγώ θα ε, το διαβιβάσω ε, και θα το συζητήσουμε και με τους συντονιστές ώστε να ληφθεί μια συγκεκριμένη απόφαση. Ωραία. Οπότε όλα καλά. Τελειώσαμε και το θέμα για αυτή την αποστολή. Θα είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το ταξίδι. Μετά, επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, έχουμε τον συνάδελφο Χριστοφόρου, που είναι ο εισηγητής μας για την ειδική έκθεση «Απαλλαγή 2019» υπαριθμών 16-2019, Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Οικονομική Λογαριασμή, υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τη χρησιμότητάς τους για τους υπεύθυνου χαράξη πολιτικής. Έχουμε μαζί μας και τον, το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Ζωάου Φιγκεραϊδο, ναι, πίσω κάθονται περισσότεροι σήμερα από ότι εδώ στα μπροστινά Να Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Οπότε σας ε, δίνω τον λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και σας ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση του ελεγκτικού συνεδρίου για να σας παρουσιάσει ε, συντομή αυτή την έκθεση του ελεγχού. Η έκθεση που σας παρουσιάζω αφορά τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς και θα ήθελα να σας τα πω σύντομα με τα βασικά ζητήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί έγινε αυτός ο έλεγχος. Και το πρώτο που θα είχαμε να πούμε από αυτού είναι ότι οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί είναι πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για περιβαλλοντικές πολιτικές, όπως για παράδειγμα οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης και η παρακολούθησή τους και το έβδομο ο ε, σχέδιο δράσης για το περιβάλλον. Είναι επικαιροποιημένε και αξιόπιστες πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές για την παρακολούθηση της Οικονομικής, Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής προέδρου για την βιώσιμη ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Οικονομική λογαριασμοί είναι ένα στατιστικό πλαίσιο που περιγράφει τους σχέσεις μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομίας. Και μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα και η συνάφεια αυτών των λογαριασμών είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο έχει σχέση με ζωτική σημασία πληροφορία ε, για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να δείξω και να σας επιστήσω την προσοχή είναι το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης αυτών των λογαριασμών. Ποιοι είναι οι κανόνες και ποιες οι ευθύνες των διαφόρων ενδιαφερομένων. Πρόκειται για ένα σύστημα πληροφοριών που περιλαμβάνει και τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη ε, τα στοιχεία, υποβάλλουν τα στοιχεία εντός των προθεσμιών και κάνουν και μία έκθεση για την ποιότητα των δεδομένων. Στη συνέχεια, μετά τα κράτη-μέλη, έχουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο της Eurostat που συλλέγει τα δεδομένα, δίνει στοιχεία για τη μεθοδολογία, αξιολογεί την ποιότητα των στοιχείων, καταρτίζει εκθέσεις και ε, προωθεί και συντονίζει πιλωτικές μελέτες. Πρόκειται για ένα σύστημα, ένα πλαίσιο στατιστικών πληροφοριών με τη συμμετοχή των κρατών μελών, τις Εθνικές Αρχές και φυσικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι ζητήσαμε εμείς και πώς θέσαμε τα ερωτήματά μας σε αυτόν τον έλεγχο. Το βασικό ερώτημα ήταν αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύστησε, διαχειρίστηκε και ε, χρησιμοποίησε σωστά τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Αυτό ήταν το βασικό ερώτημα. Και προκειμένου να λάβουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αξιολογήσαμε πώς ε, ε, διαχειρίστηκε την ανάπτυξη αυτών των λογαριασμών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν κάλυψαν τις ανάγκες των ηθινόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα σας πω εν συντομία ποια είναι τα πορίσματά μας. Το στατιστικό πλαίσιο για τους ε, ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς μέχρι τώρα δεν ε, έχει κατορθώσει να είναι πλήρες. Και στο συμπέρασμα αυτό καταλήξαμε διότι διαπιστώσαμε ότι μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ένα σύνολο περιβαλλοντικών λογαριασμών που να καλύπτουν τις ανάγκες. Δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο το οποίο καθορίζει τις ανάγκες και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες δεδομένων για τους ε, πολιτικούς ηθήνοντες και την παρακολούθηση. Και οι ανάγκες αυτών των περιβαλλοντικών λογαριασμών δεν είναι πουθενά σαφώς εκπεφρασμένες και δεν υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για χάραξη πολιτικής και παρακολούθηση. Η στρατηγική δεν συμπληρώθηκε και από ένα πλήρες σχέδιο δράσης. Υπάρχει μια στρατηγική για τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς λογαριασμούς, αλλά δεν υπάρχει ένα διεξοδικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των στόχων υπάρχουν διαδοχικές στρατηγικές οι οποίες επαναλαμβάνουν κάποιους βασικούς στρατηγικούς στόχους ε, για πάνω από μια δεκαετία. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν επίσης και κάποιες ελλείψεις που διαπιστώσαμε στον έλεγχό μας. Ελλείψεις κατά την εφαρμογή των περιβαλλοντικών λογαριασμών που σημαίνει ότι δεν ήταν τόσο σχετική με τη χάραξη πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφάρμοσε αυτά τα μοντέλα λογαριασμών χωρίς μια πλήρη ανάλυση κόστους ωφελίας. Και η εφαρμογή των μοντέλων περιβαλλοντικών λογαριασμών χρειάστηκε περίπου μια δεκαετία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως διαπιστώσαμε επίσης, δεν χρησιμοποίησε τα μοντέλα αυτά σε όλες τις σχετικές πολιτικές. Παραδείγματος χάρη δεν χρησιμοποιούνται στις πλήρες δυνατότητες τους για την παρακολούθηση πολιτικών, κυρίως την παρακολούθηση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και το 7ο περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης και αυτά τα μοντέλα των ε, ε, λογαριασμών δημοσιεύονται ξεχωριστά, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική εικόνα ε, με εναλλακτικέ πηγές δεδομένων που μας επιτρέπουν να έχουμε και μια συνολική εικόνα. Τα τελικά μας πορίσματα αφορούν προκλήσεις για την έγκαιρη συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων. Όσον αφορά στις προκλήσεις ε, για τη συλλογή δεδομένων, διαπιστώσαμε ότι κάποια από τα δεδομένα που δημοσιεύονται, δημοσιεύονται πιο γρήγορα από ό,τι απαιτείται, αλλά ε, δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι δυνατότητες για πιο έγκαιρη παροχή δεδομένων. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ε, δεν επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν πότε είναι ε, διαθέσιμα κάποια δεδομένα. Επίσης υπάρχουν κάποιες προκλήσεις ως προς την ποιότητα των δεδομένων. Τα κράτη-μέλη έδωσαν δεδομένα τα οποία δεν συνοδεύονταν και από αρκές πληροφορίες ώστε η Eurostat να αξιολογήσει καταλήλως την ε, ποιότητα των δεδομένων. Η Eurostat επίλυσε τα προβλήματα τα οποία έθετε το κάθε κράτος μέλος, αλλά κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για μεθοδολογικά προβλήματα ε, αναπτύσσονται ε, σε πορεία ετών και επομένω μπορεί να αποτελούν και πρόσκομα για τα ποιοτικά δεδομένα. Κάνουμε λοιπόν τρεις συστάσεις ε, κατ' ουσίαν. Η πρώτη είναι ένα στρατηγικό πλαίσιο για τα δεδομένα περιβαλλοντικών λογαριασμών, το οποίο θα είναι ενισχυμένο. Το δεύτερο αφορά το κατά πόσον τα μοντέλα για τη χάραξη πολιτικής είναι αυτά που χρειαζόμαστε και η τρίτη σύσταση είναι να είναι έγκαιρα αυτά τα δεδομένα για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμού, να δίνονται γέρο. Πρέπει να πω, κυρία Πρόεδρε και αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ότι εμείς θεωρούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από αυτόν τον έλεγχο, διότι καταφέραμε να έχουμε μια πλήρη ε, και ειλικρινή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να πω ότι είμαστε και πολύ ικανοποιημένοι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχθηκε πάρα πολλές από τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις μας. Ε, είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που είχαμε και με τα τελικά αποτελέσματα αυτής της δουλειάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα δεν ξέρω να σας ρωτήσω, θα τοποθετηθεί πρώτα η Κομισιόν ή εσείς ως εισηγητής. What do you wish? Θέλετε. To... Να θέλει η Κομισιόν. Ωραία. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Κομισιόν και μετά εσείς. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Βίρτς. Ευχαριστώ. κυρια Πρόεδρε, θα μιλήσω αγγλικά. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλατε το θέμα αυτό στην μέση τα Ευχαριστώ και το ελεκτικό συνέδριο. Σας ευχαριστώ για την έκθεση και την ειλικρινή συνεργασία. Ε, ήταν σαφές ε, κατά τη διάρκεια του ελέγχου πως γνωρίζαμε τις ελλείψεις που επισημάνατε στα ευρήματα και συνεχίζεται η δουλειά. Οπότε δεχόμαστε όλες τις συστάσεις που κάνετε για να βελτιωθεί το στατιστικό πλαίσιο, η σημασία των λογαριασμών για να μπορούν να είναι και χρήσιμοι και βεβαίως το έγκαιρο των δεδομένων. Να σας πω λοιπόν ποια είναι τα σχέδιά μας. Ήδη πέρσι πριν από τον έλεγχο προετοιμάζαμε την επόμενη στρατηγική για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς. Τα είχαμε συζητήσει με τα κράτη-μέλη. Αναφέρατε πως η Eurostat παίρνει τα δεδομένα, αλλά τα εθνικά στατιστικά συστήματα μας δίνουν τα δεδομένα αυτά και μαζί αποφασίζουμε για τη στρατηγική για τα επόμενα χρόνια. Και μετά, όσο γινόταν ο έλεγχος, προετοιμάζαμε το σχέδιο εφαρμογής. Αναφέρατε ότι δεν υπήρχε σαφές σχέδιο δράσης. Έχουμε ήδη συζητήσει με τους ειδικού στα κράτη-μέλη την εφαρμογή και αν και το σχέδιο δράσης υπήρχε. Τώρα στην εφαρμογή θα δώσουμε προτεραιότητα σε δράσεις για να, ε, όπως είπα, έχουν μεγαλύτερη συνάφεια οι λογαριασμοί και θα θέσουμε συγκεκριμένους στόχους και εκτιμήσεις προϋπολογισμού. Έχουμε προβλέψει και μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση που θα ξεκινήσει για το επόμενο σχέδιο δράσης μέχρι το 2022 ε, για να δούμε τις συστάσεις που κάνατε. Να αναπτύξουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και τις αναγκές δεδομένων, την διάδοση των δεδομένων έτσι ώστε οι χρήστες μας να τα γνωρίζουν, να γνωρίζουν εγκαίρως πότε θα τα δημοσιεύσουμε Αναφέρατε επίσης πως ε, οι λογαριασμοί δεν ε, συνδέονται. Υπάρχουν διάφορα στοιχεία στους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς που δεν συνδέονται. Συνολικά θα ήθελα να πω πως οι λογαριασμοί αυτοί, κάθε κομμάτι τους, ε, περιλαμβάνει διάφορα στατιστικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα και παρουσιάζει τα δεδομένα σε ένα πλαίσιο και δείχνει πώς συνδέονται οι πληροφορίες. Αυτό θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να ακούσω και το κοινοβούλιο και αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και άλλες διευκρινήσεις. Ευχαριστώ. Τώρα ο εισήγητης μας ο κ. Χριστοφόρου. Ε, πιστεύω ότι η εξέταση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οικονομικών λογαριασμών είναι μια πολύ σημαντική δραστηριότητα για όλους μας. Ε, αυτόν το Κοινοβούλιο πολλές φορές εξέφρασε την αναγκαιότητα χάραξη σημαντικών στρατηγικών για το περιβάλλον. Και αυτές οι στρατηγικές δεν πρέπει να γίνονται αυτοσκοπός. Δηλαδή, όλοι μα είμαστε υπέρ του περιβάλλοντο και πολλέ φορέ υπάρχει φοβία να διατυπώσουμε οποιασδήποτε στάσει όσον αφορά το οικονομικό κόστο ή ακόμα και τη διασπάθηση που μπορεί να γίνεται. Αναδεικνύεται μέσα από του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού οικονομικού λογαριασμού ότι μπορεί να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για να υπάρξει στενή παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι περιβαλλοντικές πολιτικές δεν είναι ανεξέλεκτες. Και θεωρώ και χαιρετίζω την εξαιρετική δουλειά που έγινε από, τον ε, αγαπητόν, ε, από το αγαπητόν εισηγητικό μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου του κ. Χουάου, αλλά ιδιαίτερα δε χαιρετίζω την θετική στάση που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί αντιλαμβάνεται ότι αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξαν σημαντικέ ελλείψει. Για μένα είναι σημαντική έλλειψη για δυναμία να μην γίνεται επακριβή, αξιόλογη, αντικειμενική ανάλυση κόστου και ωφέλου. Όπω και μέσα από του περιβαλλοντικού οικονομικού λογαριασμού μπορούμε να εντοπίζουμε όλε εκείνε τι περιπτώσει ότι υπάρχει επιβάρηση και καταστροφή του περιβάλλοντο και να αναδεικνύεται ποιο πρέπει να καταβάλει το κόστο. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν πραγματικά υιοθετεί τι εισηγήσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, σίγουρα την επόμενη χρονιά θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, αλλά αυτή η υλοποίηση να μην γίνει μόνο σε επίπεδο θεωρητικό, αλλά να γίνει σε πρακτικό. Το άλλο σημαντικό κλειδί για όλα αυτά είναι τα κράτη-μέλη. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι τα κράτη-μέλη δεν ανταποκρίνονται πλήρω και δεν παρέχουν έγκαιρα τα στοιχεία. Στοιχεία τα οποία δεν παρέχονται έγκαιρα, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά καταστρέφουν την προσπάθεια για να υπάρχει αποδοτικότητα σε αυτού του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού οικονομικού λογαριασμού. Άρα, αφού όλοι εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη, πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι θα υπάρχουν επιπτώσει εκεί και όπου υπάρχει καθυστέρηση στην διοχέδευση αυτών των στοιχείων και αυτών των αποτελεσμάτων. Εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικέ οι εισηγήσει που γίνονται από το ε, ελεκτικό συνέδριο. Αυτέ όπω γίνονται είναι όλε εφικτέ να υλοποιηθούν και οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επόμενη χρονιά να είναι εδώ απλώ για να μα πει ότι τι υλοποίησε όλε και εμεί χαιρετίζουμε το γεγονό ότι είναι θετική προ αυτή την κατεύθυνση. Όμω ταυτόχρονα θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικέ ελλείψει όσον αφορά τη στρατηγική για του περιβαλλοντολογικού λογαριασμού, ιδιαίτερα το 2019-2023, και θα πρέπει να περιγραφεί ένα διεξοδικό σχέδιο δράση για να καλύπτει τι μελλοντικέ εργασίε στην περιοχή συμπεριλαμβανομένων των οροσύμων και των εκτιμήσεων του προπολογισμού. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε ότι τα σημεία δράση προτείνονται σε ένα έγγραφο εφαρμογή, χωρί ωστόσο να καθορίζεται ο τρόπο με τον οποίο πρέπει ή οφείλουμε να τα υλοποιήσουμε αυτέ τι δράσει και χωρί να συμπεριλαμβάνονται οι ημερομηνίε στόχοι για αυτά τα σημεία. Και αυτό είναι ένα σημαντικό. Για μα, όπω είπα, είναι σημαντική η ανάδειξη του κόστου και ωφέλου. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μια πιο πλήρη πληροφόρηση και ενημέρωση, δηλαδή στο μέσο τη διαδικασία η Επιτροπή μπορεί να μα απελευθερώνει δεδομένα για την πρώτη φάση που θα αφορούν συγκεντρωτικά στοιχεία για μια δράση και στη δεύτερη φάση θα υπάρχουν τα λεπτομερέστερα. Με όλα αυτά θέλω να πω για μια ακόμη φορά ότι εμείς στηρίζουμε τις δράσεις για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, ότι είναι ένας σημαντικός τομέας που αναδεικνύεται σήμερα μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πραγματικά αποτελεί και πρόκληση ιδιαίτερα με την ε, υλοποίηση της συμφωνίας για τον Green Deal αν και αυτές οι πολιτικές, πέρα από τις πολιτικές περιβάλλοντος και βιώσιμος ανάπτυξης, εισέρθουν και αυτές μέσα στη λογική της εξέτασης, άρα εκεί πρέπει να είμαστε πιο πλήρει, πιο αποτελεσματικοί και πιο έτοιμοι να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την όλη κατάσταση έχοντας ως στόχο την διαφάνεια, έχοντας ως στόχο την εξοικονόμηση και την αύξηση της αποδικοδοτικότητας των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχοντα υπόψη μα ότι με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι πολιτικέ για το περιβάλλον και θα έχουν τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα για όλους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Κύριε Μπούγε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελεγκτικό Συνέδριο για αυτή την πολύ ε, σημαντική ε, έκθεση και να ευχαριστήσω και τον συνάδελφο τον κύριο Χριστοφόρου για το σχέδιο έκθεσης που είναι πλήρες και πολύ ισορροπημένο. Το ουσιαστικό και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, και όπως πολύ σωστά υπενθύμησε ο εισηγητής, ε, η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ανέλαβε καθήκοντα αρχές Δεκεμβρίου, θεωρεί ότι το περιβάλλον και η προστασία του πλανήτη μας είναι απόλυτη προτεραιότητα μέσω της συμφωνίας του Green Deal και του στόχου ε, της ε, ε διακοπής της χρήσης των υδρογων το 2050 και στην πρόσφατη προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ, όλοι ρωτηθήκαμε από τους πολίτες για τα θέματα αυτά ε, και περιμένουν από εμά και θα μας κρίνουν για το πώς θα καταφέρουμε συλλογικά να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όταν λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι στον τοίχο για τα θέματα αυτά και περιμένουν να κάνει κάτι, πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να δράσει ώστε να συμφουλιωθεί με τους Ευρωπαίους πολίτες ή θα τους απογοητεύσει και θα χειροτεύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λοιπόν συλλογική ευθύνη και πρέπει να την αναλάβουμε όλοι για να βελτιώσουμε τα πράγματα και ε, είναι σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένους δείκτες εύστοχου δείκτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι περιβαλλοντικοί οικονομικοί λογαριασμοί να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα προσανατολισμένοι και εστιασμένοι στην επίτευξη των στόχων μας. Η έκθεση αναφέρει πολύ καλά πώς επιλέχθηκαν τα διάφορα ε, μοντέλα και πώς αναπτύχθηκαν σε το χρόνο και ε, θα ψηφίσουμε σύντομα στην Ολομέλεια το νομοθετικό κείμενο που ε, καθορίζει ένα πλαίσιο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, όπως την έχουμε ε, αποκαλέσει. Και ο στόχος είναι όχι να δούμε μόνο τα οικονομικά κριτήρια στις επενδύσεις, αλλά φυσικά και τα οικολογικά, κοινωνικά και ε, τα κριτήρια διακυβέρνησης. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ουσιαστική πρόοδος. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να φροντίσουμε και τα εργαλεία μας αυτά να αναπτυχθούν για να καλύψουν τις ανάγκες μας. Πολύ σωστά το επισημαίνει ο εισηγητής. Ε, θα πρέπει να καθορίζουν τις ευρωπαϊκές μας πολιτικές ε, τα modules αυτά και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνεται. Και ένα στοιχείο αμφιβολίας για να ολοκληρώσω κυρία Πρόεδρε. Το ελεγκτικό συνέδριο λέει ότι κάποια κράτη-μέλη δεν δίνουν κανένα στοιχείο ακόμα χωρίς κάποιες κυρώσεις και κάποια διαδικασία επί παραβάση, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ε, διαπιστώνω κύριε Σιγητά ότι και εσείς ρωτάτε στην τελευταία παράγραφο και ζητάτε από την Κομισιόν να πιέσει τα κράτη-μέλη ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν ε, συγκρίσιμοι ορισμοί και θα μπορέσουμε να έχουμε δείκτες σε όλα τα κράτη-μέλη. Εγώ θα πήγαινα ακόμα παραπέρα εάν χρειαστεί και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε αποτελεσματικούς και συγκεκριμένους λογαριασμούς, ε, κάτι το οποίο είναι αδύνατο χωρίς εναρμονισμένα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Συμφωνώ και με τους δύο. Και εγώ εξεπλάγει όταν έμαθα ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν δίνουν δεδομένα. Και δεύτερον, ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν δίνουν έγκυρα δεδομένα ή που δίνουν δεδομένα χωρίς να δίνουν και το συγκείμενο. Ε, που δεν τα καθιστά και τελείω άχρηστα αυτά τα δεδομένα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι έγκυρα ως προς το να διαμορφωθεί μια συνολική εικόνα για το πώς έχουν τα πράγματα. Δεύτερο πράγμα που με εξέπληξε είναι το γεγονό ότι ενώ γίνονται συζητήσει εδώ και καιρό για την Πράσινη Συμφωνία, εξακολουθούμε να μην έχουμε μια, δεν, να μην έχουμε μια συνολική εικόνα μέσω των δεδομένων, ε, γιατί ακριβώ τα δεδομένα που αυτή τη στιγμή έχουμε στη διάθεσή μα δεν είναι έγκυρα. Από αυτή την άποψη ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για το γεγονός ότι μας επέστησε την προσοχή μας σε αυτό το θέμα γιατί το επόμενο διάστημα βεβαίως θα, θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε διάφορες νομικές πράξεις γύρω από το περιβάλλον και ε, βεβαίως θα είναι ύψης της σημασίας να έχουμε πολύτιμα και αξιόπιστα δεδομένα γιατί ε, δεν είναι μόνο κάτι που μας ε, αφορά εδώ ως ε, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, χρειάζεται όλα αυτά τα δεδομένα και να συλλέγονται με έναν ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο, ώστε να είναι και συγκρίσιμα για να μπορούν να ε, αξιοποιηθούν στο πλαίσιο μιας συνολικής εικόνας που θέλουμε να σκιαγραφίσουμε και να διαμορφώσουμε. Η Κομισιόν ίσως θα ήθελε να μας ενημερώσει ποια είναι τα κράτη-μέλη, πόσα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία δεν υποβάλλουν δεδομένα και ποια μέτρα έχει πάρει μέχρι στιγμής η Κομισιόν για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Ναι. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξη που επιδεικνύεται για τους, για τους περιβαλλοντικούς λογαριασμούς και την ε, ε, ανάγκη να υπάρχουν δεδομένα και για τη δικιά σας δουλειά. Για το ερώτημά σας πόσα κράτη-μέλη δεν έχουν υποβάλει δεδομένα, έχουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα με τρία κράτη-μέλη συγκεκριμένα. Χρησιμοποιούμε όλα τα νομικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Κάνουμε δηλαδή αξιολογήσεις συμμόρφωσης. Δίνουμε και βοήθεια στα κράτη-μέλη αυτά για τους ελέγχους που προβλέπονται από τον κανονισμό, για νέα προγράμματα με πιλωτικά προγράμματα και υποστηρίζουμε τα τρία αυτά κράτη που είναι και ε, τα μικρότερα κράτη που δεν έχουν τα τεχνικά μέσα. Για αυτά τα κράτη-μέλη ε, κάνουμε ε, βάσιμες αξιολογήσεις για την ε, για την ε, κατάρτιση τέτοιων λογαριασμών. Βεβαίω, για τη δική σα δουλειά χρειάζονται εθνικοί λογαριασμοί. Εμεί έχουμε και περιφερειακού λογαριασμού. Του αξιοποιούμε ω τι πληροφορίε των κρατών μελών για να μπορούμε να καταρτήσουμε αυτού του ευρωπαϊκού λογαριασμού για να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνουν είναι αξιόπιστα με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε. Χρησιμοποιούμε και αξιοποιούμε ό,τι έχουμε στη διάθεσή μα. Όμω είναι αλήθεια ότι με την Πράσινη Συμφωνία και την περιβαλλοντική διάσταση των θεμάτων να λαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη σημασία είναι πραγματικά πολύ σημαντικέ οι συστάσει, αυτές που μα επέβαλε το ελληνικό συνέδριο και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να τις εφαρμόσουμε. Τα δεδομένα αυτά, ρωτάει η πρόεδρο, είναι αξιόπιστα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε και το ε, ε, ελεγκτικό συνέδριο. Η αξιοπιστία των, των δεδομένων είναι αυτή που μας ενδιαφέρει, γιατί πολλές φορές συλλέγονται σε περιφερειακό επίπεδο, ξέρουμε ότι εκεί τα συστήματα μέτρησης και συλλογής δεδομένων είναι διαφορετικά. Οπότε τα δεδομένα που καταλήγουν εδώ σε εμά είναι τελικά έγκαιρα και αν είναι σε ποιο βαθμό. Να ξαναδώσω το λόγο στην Κομισιόν και στο Ελληνικό Συνέδριο. Ναι, τα δεδομένα που έχουμε είναι αξιόπιστα. Θα μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε περισσότερα δεδομένα, θα μπορούσαν να υποβάλλονται πιο έγκαιρα, όμως τα δεδομένα που τελικά καταλήγουν σε εμά είναι και έγκυρα και συγκρίσιμα. Δεν ξέρω ότι και στη χώρα μου υπήρξαν κάποια προβλήματα στο πρόσφατο παρελθόν, οπότε ε, με, με, ανησυχεί λίγο αυτή η απόλυτη δήλωσή σας, γιατί στην Ευρώπη ποτέ δεν είναι όλα τα δεδομένα έγκυρα και αξιόπιστα. Ποτέ δεν, δεν μου έχει ξανασυμβεί. Ωραία το θέσατε, αλλά να σας πω την αλήθεια δεν με πείθετε και 100%. Να δούμε λίγο τι θα μας πει και το ελληνικό συνέδριο. Για την εγκυρότητα των δεδομένων και την αξιοπιστία τους. Μπορείτε να μας πείτε κι εσείς δύο λόγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, ε, θα ήθελα να κάνω και κάποια άλλα σχόλια ε, έπειτα από τις παρεμβάσεις των βουλευτών και τις απαντήσεις που ακούσαμε από την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Χριστοφόρου, για την εξαιρετικά ολοκληρωμένη ε, έκθεση που έχει συντάξει για την ειδική έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Οι υπερβολητικοί λογαριασμοί είναι πραγματικά σημαντικότατο εργαλείο για την παρακολούθηση διαφόρων πολιτικών που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό είναι και το βασικό σημείο ε, από πολιτικής ε, άποψης. Και όπως είπε και ο κύριος Μποαγιέ, είναι πολύ σημαντικό επίσης και για το μέλλον, γιατί σχετίζεται και με τη Νέα Πράσινη Συμφωνία. Και θα είναι, θα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών που θα συμπεριλαμβάνονται στην ε, Πράσινη Συμφωνία. Θα ήθελα να απαντήσω και στην ερώτηση που έθεσε ο κ. Μπουαγέ. Όσον αφορά την καθυστέρηση των κρατών μελών στην αποστολή των δεδομένων διότι όπως σας είπα στην έκθεσή μας έχετε ε, στοιχεία στον πίνακα 3 για τα θέματα αυτά και επίσης και στην παράγραφο 50. Υπάρχουν πληροφορίες επ' αυτού, αλλά και κάποια θέματα τα οποία απάντησε ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα επίσης ε, και να απαντήσω στην ερώτηση της Προέδρου. Σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών. Όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, εμείς ισχυριζόμαστε ή μάλλον επιστούμε την προσοχή σας στην, έκθεση, στην παράγραφο 52 της έκθεσής μας. Θεωρούμε ότι η Eurostat πρέπει να ζητά περισσότερες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δεδομένων που αποστέλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, όσον αφορά τις ερωτήσεις που ακούστηκαν σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνει η Κομισιόν απέναντι στα κράτη-μέλη που δεν απαντούν έγκαιρα και σωστά και εκεί υπάρχουν κάποια στοιχεία στην ε, έκθεσή μας. Υπάρχει για παράδειγμα σύσταση 3 όπου λέμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αξιοποιεί τα ήδη διαθέσιμα εργαλεία για να βελτιωθεί το έγκαιρο τη υποβολή των στοιχείων από τα κράτη-μέλη. Η Κομισιόν έχει ήδη διάφορα εργαλεία στα χέρια τη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα κράτη-μέλη απαντούν και υποβάλλουν τα δεδομένα έγκαιρα και ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι σωστά. Α, να πω επίση ότι οι συστάσει του συνεδρίου στην έκθεση αυτή αποτελούν κοινό αποτέλεσμα της συνεργασίας της δικής μας με τις υπηρεσίες κομισιών. Υπάρχει συναντήληψη όσον αφορά τις αδυναμίες των συστημάτων. Γι' αυτό και θα μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι κάνει ήδη η Κομισιόν στην κατεύθυνση της εφαρμογής των συστάσεων στις οποίες, όπως είπα, καταλήξαμε μαζί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι βέβαιο ότι θα το ξαναδούμε το θέμα αυτό. Ε, ο εισηγητής μας ο Λευτέρης Χριστοφόρου μήπως θέλει το λόγο έτσι, για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ότι ο στόχος όλων μας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ε, Ελεκτικού Συνεδρίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εμέναν του εισηγητή αλλά και του αγαπητού συνάδελφου του βοηθού εισηγητή είναι κοινό. Αφενό με να στηρίξουμε τι περιβαλλοντικέ δράσει και αφετέρου όμω αυτέ οι δράσει να μην είναι ανεξέλεκτε. Οικονομία και περιβάλλον πάνε μαζί. Και πιστεύω ότι ιδιαίτερα πρέπει για τα πάντα πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει ανάλυση κόστου και ωφέλου. Δεν μπορεί να γίνονται ανεξέλεκτα στο βωμό τάχατε μια περιβαλλοντική ε, συνείδηση ή μια περιβαλλοντική πολιτική. Άρα πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να εργαστούμε και να πετύχουμε του στόχου που δεν πετύχαμε μέχρι σήμερα και χαιρετίζω ξανά και την προθυμία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την εξαιρετική εργασία που έγιναν από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Και εγώ σα ευχαριστώ και του τρει. Τον εισηγητή, την Κομισιόν και το Ελληνικό Συνέδριο. Σα ευχαριστώ θερμότατα. Και ήρθε νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν και ο συνάδελφος Φλάναγκαν. Προχωρήσαμε γρήγορα. Κάτι που μας δίνει τη δυνατότητα να περάσουμε στο σημείο 5 τη ημερήσια διάταξη, η ειδική έκθεση σταθεροποίηση του εισοδήματο των γεωργών, ολοκληρωμένη μένει η εργαλειοθήκη. Όμω πρέπει να αντιμετωπιστούν η ανεπρική ε, αξιοποίηση ορισμένων μέσων και η υπεραντιστάθμιση. Θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στο μέλο του Ελληνικού Συνεδρίου, τον κύριο Σάμο Γέρεπ, για να μα παρουσιάσει την ειδική αυτή έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω σήμερα την ε, πιο πρόσφατη έκθεση για το μέσο σταθεροποίησης του εισοδήματο των Γεωργών. Θα σας παρουσιάσω τα απορίσματά μας και τις συστάσεις μας, ιδίως αυτά που δεν έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάσαμε αν είναι πλήρη και συνοπτικό το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων και όπου είχαμε εργαστία, εργαλεία τέτοια που χρησιμοποίησαμε, είδαμε αν ήταν αποτελεσματική η εφαρμογή και είχαμε στήριξη για ασφάλιση και εξαιρετικά μέτρα μετά από την ε, ρωσική ε, απαγόρευση, το ρωσικό εμπάργκο το 2014. Να σα παρουσιάσω συντομία τα πορίσματά μα. Όσον αφορά τη ε, μέσα διαχείριση κινδύνων, κινδύνου διαπιστώσαμε ότι η χρήση της ευρωπαϊκής στήριξης είναι χαμηλή. 17 κράτη-μέλη δεν εφάρμοσαν αυτή τη στήριξη όπως δείχνει ο χάρτης. Πάνω από το 90% των σχεδιαζόμενων ευρωπαϊκών δαπανών είναι για ασφάλιση ε, το υπόλοιπο είναι και για το εργαλείο σταθεροποίησης ε, και είχαμε λιγότερο από 8% των ε, ασφαλισμένων γεωργών που στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του πυλώνα 2. Για τα δύο κράτη-μέλη που έχουμε ευρωπαϊκή ασφάλιση, η Ιταλία και τη Γαλλία, ένα μεγάλο ποσοστό είναι στον τομέα του ίνου. Αυτό σχετίζεται και με το κίνδυνο μόχλευσης. Περίπου 41 δις το χρόνο άμεσες ενισχύσεις διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην στρατηγική διαχείριση κινδύνου. Όσο μεγαλύτερο είναι το μερίδιο άμεσων ενισχύσεων στο γεωργικό εισόδημα, τόσο χαμηλότερη είναι η χρήση ασφάλισης και αντιστρόφως. Επίσης, οι άμεσες ενισχύσεις ε, ε, βοηθούν ε, την ανθεκτικότητα των γεωργούν με δύο τρόπους. Είναι και επιπλέον εισόδημα, αλλά βοηθούν και τους γεωργούς μέσω διαφόρων περιβαλλοντικών απαιτήσεων υπό την προπόθεση ότι θα αλλάξουν τη συμπεριφορά του και έτσι θα βελτιώσουν την ανθεκτικότητά τους. Τώρα εφαρμόζονται μέσω του γκρίνου και στο μέλλον ε, μέσω τη ε, τη της αμύψης Αυτό θεωρήθηκε και ότι είναι και το πιο σημαντικό προληπτικό μέτρο ε, στην ε, Γεωργία. Κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ε, είναι λίγο αντιφατικά ως προς τα κίνητρα που παρέχουν. Κάποια εξαιρετικά μέτρα χρησιμοποιήθηκαν ε, για συγκεκριμένους κλιματικούς κινδύνους. Αυτό δεν θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική χρήση μέσων, όπως για παράδειγμα την ασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι ασφαλισμένοι γεωργοί δεν μπορούν να υποφαληθούν εξαιρετικών μέτρων και αυτό φυσικά τους αποθαρρύνει από το να ε, συνάψουν μια, μια ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης, ε, τα οποία μπορεί να αποθαρρύνουν βεβαίως τους γεωργούς και να μην ασφαλιστούν, διότι θεωρούν ότι θα μπορούσαν να αποφαληθούν από μέτρα τα οποία λαμβάνονται εκ των υστέρων. Η ασφάλεια και τα αμοιβαία κεφάλαια είναι συμπληρωματικά μόνο όταν αντιμετωπίζουν διαφορετικούς κινδύνους. Τα κράτη-μέλη συλλέγουν πληροφορίες για τα προγράμματα διαχείρισης κινδύνου που δεν συλλέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποιοι δείκτες παραγωγής όσον αφορά το ε, κεφάλαιο το οποίο ασφαλίζεται ή οι εκτάσεις που ασφαλίζονται συλλέγονται από τα κράτη-μέλη όπως για παράδειγμα από τη Γαλλία και την Ιταλία ενώ η Κομισιόν δεν συλλέγει τέτοια στοιχεία για να έχει εικόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα δείκτη αποτελεσμάτων, ποσοστό των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχει σε προγράμματα διαχείριση ε, κινδύνου, είναι ένα πάρα πολύ αμφίσιμο δείκτη που δεν μα επιτρέπει να κάνουμε και σύγκριση μεταξύ κρατών μελών. Τώρα θα επικεντρωθώ σε κάποια απορίσματα όσον αφορά τα εξαιρετικά μέτρα τα οποία δόθηκαν για τον τομέα των οποροκυπευτικών ε, μετά από το ρωσικό εμπάργο το 2014. Είχαμε περίπου 413 εκατομμύρια ευρώ από τις ευρωπαϊκές δαπάνες. Ε, δεν υπήρχαν συγκεκριμένα κριτήρια για να εξεταστεί η χρήση τέτοιων εξαιρετικών μέτρων. Το μεγαλύτερο μέρο τη στήριξη πήγε στην παραγωγή των μήλων για ποσότητε οι οποίε αποσύρθηκαν και υπήρξε και η στήριξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά το ρωσικό εμπάργκο, αυξήθηκαν οι εξαγωγέ μήλων και σε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, που σημαίνει ότι κάποιε άλλε αγορέ εκτό Ρωσία βρέθηκαν για την εξαγωγή. Αυξήθηκαν συνεχώς οι εξαγωγές ε, από το 2014 και μετά. Το 2009 όμως δεν είχαμε εκτακτά μέτρα. Τα εξαιρετικά μέτρα ε, αυτά ελήφθησαν για τέσσερα χρόνια και καταλήξαμε το συμπέρασμα ότι χρησιμοποιήθηκαν και για ε, προγράμματα ε, διαρθρωτικών πλεονασμάτων σε ροδάκινα και νεκταρίνια και είδαμε την παραγωγή μέχρι το 2017 και είδαμε ότι χρησιμοποιήθηκαν και για αυτά. Υπήρχαν επίση κάποιε περιπτώσει που δόθηκαν υπερβολικέ αποζημιώσει, δηλαδή η ευρωπαϊκή στήριξη για απόσυρση μήλων από την αγορά ήταν υψηλότερη από την τιμή αγορά. Αυτά σημαίνει ότι το μέτρο είναι ιδιαίτερα δελεαστικό. Καταλήξαμε ότι το κόστος ε, των ε, προγραμμάτων απόσυρσης ήταν πολύ ψηλό. Ε, μπόρεσε να γίνει και επεξεργασία σε χυμό για κάποια προϊόντα τα οποία αποσύρθηκαν από την αγορά και διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ψηλήρισε, πλήρωσε ακριβά τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια για χυμό. Ένα λίτρο χυμό ε, για κατανάλωση από άτομα που έχουν ανάγκη ήταν κόστος 4,25 ευρώ, τετραπλάσιο του κόστους ενός χυμού στα σούπερ μάρκετ. Και επειδή πληρώθηκαν ε, ε, σε είδο όσοι κάνουν την πεταποίηση, πολλά από τα προϊόντα ξαναβρέθηκαν στην αγορά και τελικά δεν δόθηκαν σε άτομα τα οποία είχαν ανάγκε. Ε, κάναμε αρκετέ συστάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα διαχείριση κινδύνου, συστήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενθαρρύνει του παραγωγού να προετοιμάζονται καλύτερα για κρίσει για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να δίνονται μέτρα για ε, πρόληψη ε, και παρεμβάσεις για να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο ανθεκτικοί οι γεωργοί. Θα πρέπει επίσης να δίνεται στήριξη για γεωργικές πρακτικές που μειώνουν την έκθεση σε κίνδυνο και μετριάζουν τους κινδύνους, τις ε, ζημίες. Συγγνώμη. Πρέπει να υπάρχει καλύτερο σχεδιασμό και παρακολούθηση τη στήριξη για ασφάλιση, ιδιαίτερα επειδή είναι χαμηλό το ποσοστό των ασφαλισμένων και το γεγονό ότι συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένου τομεί και σε μεγαλύτερου παραγωγού. σω λοιπόν υπάρχει προστιθέμενη αξία εδώ για την ε, ε, ε, ασφάλιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν είναι και η βέλτιστη στιγμή να δούμε την ε, στήριξη αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι κατάλληλη επιχειρηματολογία αυτή, διότι θα μπορούσαμε να το έχουμε στα νέα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου που ξεκινούν το 2021 και θα έχουμε την ε, προστιθέμενη αξία που είναι ένας από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης που θα πρέπει να εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα μέτρα. Η επόμενη σύσταση ήταν να παρακολουθούνται οι δαπάνες μέσω συγκεκριμένων ενδεικτών, όπως για παράδειγμα έκταση και κεφάλαιο που ασφαλίζεται, που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο κράτου μέλους και να υπάρχουν κατάλληλοι δείκτες γι' αυτό. Όσον αφορά τα εξαιρετικά μέτρα, συστήσαμε ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκρινίσει τα κριτήρια για την ε, έναρξη και τη λήξη των εξτάκτων μέτρων και να υποστηρίξουμε τη χρήση τέτοιων εκτάκτων μέτρων για εξαιρετικά καιρικά φαινόμενα, για γεωργούς που έχουν χρησιμοποιήσει μέτρα διαχείρισης κινδύνων και έχουν δοθεί ε, και κατάλληλα μέτρα στους γεωργούς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι είναι εύστοχη αυτή η σύσταση, αλλά θέλει να έχει τη διακριτική ευχαίρεια να παρέμβει αναπερίπτωση όταν έχουμε εκτακτά μέτρα. Ωστόσο, εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνει η σύσταση αυτή, γιατί αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται ήδη σε αρκετά κράτη-μέλη και έχουμε ένα σύστημα το οποίο βασίζεται σε εύρωστα κριτήρια, γιατί έτσι μπορούμε να δείξουμε και στους γεωργού εκ των προτέρων ότι έκτατα μέτρα για ακραία καιρικά φαινόμενα εφαρμόζονται μόνο όταν είναι αιτιολογημένο. Επίσης, ε, συνήθως μετά από καταστροφικά γεγονότα, ε, ε, εάν δοθούν αμέσως έκτακτα μέτρα, οι γεωργοί δεν έχουν κίνητρο να μετριάσουν τους κινδύνους. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ε, προσαρμογή της αποζημίωσης για επιχειρήσεις απόσυρσης προϊόντων, ώστε να μην είναι εις βάρος των τιμών αγοράς ε, στα κράτη-μέλη ε, της παραγωγής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται αυτή τη σύσταση γιατί σημαίνει ότι δεν θα έχουν δυνατότητα να παρέμβουν σε κρίσεις αναπερίπτωση. Εμείς παραμένουμε σε αυτή τη ε, σύσταση διότι πρέπει να έχουμε εκ των προτέρων υπολογισμό για να έχουμε ισότιμη μεταχείριση των γεωργών σε αντίστοιχε περιπτώσει. Στοιχεία για τι τιμέ τη αγορά είναι διαθέσιμα στα κράτη-μέλη και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ελέγξουν ότι η στήριξη για την απόσυρση δεν είναι υψηλότερη τη τιμή αγορά και δεν έχουμε υπερβολική αποζημίωση. Επίσης θα πρέπει να αξιολογήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι πρακτικό να έχουμε ποσά κάτω από το 100% και ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βοηθήσουν εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ελπίζω να βοήθησα να διευκρινίσουμε και τις ε, διαφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις συστάσεις αυτές και με στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Θα θέσω και στον κύριο Φλάναγκαν το ίδιο ερώτημα που έθεσα και στον κύριο Χριστοφόρο. Να ακούσουμε πρώτα την ε, Κομισιόν για να μιλήσετε εσείς μετά ή πρώτα εσάς. Ε, Κομισιόν. Κομισιόν ή εσείς, τι θέλετε. Ναι, ναι, ας ακούσουμε την Κομισιόν. Ωραία. μια που ακούσαμε ότι υπάρχουν κάποιες ε, διαφορές απόψεων ε, με το ελεκτρικό συνέδριο. Περιμένω να ακούσω τι έχετε να πείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι έχουμε κάποιες ε, διαφορές απόψεων, αλλά αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την αξία της έκθεσης, η οποία είναι επίκαιρη και χρήσιμη. Και είναι χρήσιμο ακριβώς να ελέγχει τα συστήματα, το ελεγκτικό συνέδριο για να δει εάν μπορούν να βελτιωθούν. Άλλο βεβαίως, για να δούμε και το τι γίνεται στους ελέγχους στα μέτρα στήριξης αγοράς και τα έκτακτα μέτρα και όπως είπε και το ίδιο το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή έχουμε τις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ που είναι άλλη μια ευκαιρία για να λάβουμε υπόψη αυτά τα ευρήματα. Οπότε σημειώσαμε την έκθεση και θα εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα που προτείνουν οι συστάσεις αν και δεχόμαστε ότι αποκλίνουμε σε κάποια σημεία. Αλλά δεν πρέπει να υπερτονίζουμε τις διαφορές ελεγκτικού συνεδρίου και κομισιών γιατί το συνέδριο αναγνωρίζει ότι αυξάνει την ανθεκτικότητα των αγροτών η κοινή αγροτική πολιτική και το καλύτερο παράδειγμα είναι το σύστημα άμεσων πληρωμών που έχει σημαντικό αντίκτυπο στην σταθεροποίηση του εισοδήματος των αγροτών που τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν καλύτερα την χαμηλότερη παραγωγή ή τις χαμηλότερες τιμές και μιλάμε για 40 δισεκατομμύρια το έτος. Ε, πολύ σημαντικό ποσό. Επίσης η Κομισιόν αναγνωρίζει την ε, σημασία των κατάλληλων εργαλείων ε, για να διαχειριστούμε κινδύνους και κρίσεις, ειδικά στον τομέα της γεωργίας που από τη φύση του είναι ιδιαίτερος ευπαθής παραδείγματος χάρη σε διάφορες επιδημίες, στον καιρό, διαταράξει του εμπορίου και άρα κυμαίνονται τα εισοδήματα των αγροτών και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αυτές τις διακυμάνσει. και η ΚΑΠ τους δίνει αυτή τη δυνατότητα μέσω της εισοδηματικής στήριξης ε, των μέτρων αγοράς, ε, εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και επενδύσεις με βάση το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και όπως είπε και το δικαστήριο Άρα γνωρίζουμε πως τα διαφορετικά μέσα που έχει η ΚΑΠΑ αναλόγως με το πως χρησιμοποιούνται μπορούν να ενισχύσουν το ένα το άλλο και βεβαίως καμιά φορά έχουν και κάποιες ε, παρενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν συνδυαστικά να λειτουργούν καλά. Και έτσι ερχόμαστε στην πρώτη σύσταση του δικαστηρίου που λέει να ενθαρρύνουμε τους αγρότες να προετοιμαστούν καλύτερα για τις κρίσεις. Η Κομισιόν τονίζει ότι οι προτάσει μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ πηγαίνουν προ αυτήν την κατεύθυνση ακριβώ. Για να διασφαλίσουμε ότι οι αγρότε θα προστατεύονται στο μέτρο του δυνατού ε, κατά τον... Ε, ραγδαίων διακυμάνσεων του εισοδήματό τους. Και βεβαίω τα κράτη-μέλη θα ωφεληθούν από το στρατηγικό σχεδιασμό επιπλέον ευελιξία ειδικά με βάση τη νέα προσέγγιση που βασίζεται στην απόδοση. Έχουμε δηλαδή ένα μοντέλο που θα μας πάει πιο πολύ στην απόδοση παρά στη συμμόρφωση. Επιπλέον, η Κομισιόν προτείνει τα εργαλεία διαχείρισης του κινδύνου να γίνουν υποχρεωτικά για τα κράτη-μέλη. Και αυτό περιλαμβάνει και τις ε, συνεισφορές στα ασφάλιστρα και βεβαίως ε, βοήθεια στους αγρότες για να αντιμετωπίσουν κινδύνους ή τις συνέπειες. Σε σχέση με τη δεύτερη σύσταση, καλύτερο σχεδιασμό και στήριξη στον τομέα των ασφαλιών, τονίζουμε ότι τα νέα εργαλεία όπως αυτά της διαχείρισης κινδύνου απαιτούν χρόνο και όσον αφορά τις δυνατότητες των εθνικών διοικήσεων αλλά και για την ενημέρωση των αγροτών. Και ε, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε ποτέ σε κάποια κατάσταση όπου το 100% των αγροτών ε, θα εκμεταλλευτούν ε, τους χάρη τα ασφάλιστρα ή τα αμοιβαία κεφάλαια. Υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον πίνακας που τονίζει ότι αρκετοί αγρότες ε, δεν ενδιαφέρονται για ασφάλειες, κάνουν τις δικές τους προβλέψεις και έχουν άλλα μέτρα μείωσης του κινδύνου. Τώρα στι προετοιμασίε για τη μελλοντική ΚΑΠ. αυτές οι πτυχές έχουν ήδη αξιολογηθεί σε πολλές εξωτερικές μελέτες και προφανώς δεν είναι μυστικό ότι τα τελευταία 20-30 χρόνια ένα μόνιμο ζήτημα είναι το πώς θα μπορούσαν οι αγρότες να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα μέσω ασφαλιών ή αμοιβαίων κεφαλαίων για να μην χρειάζονται μέτρα στήριξης αγοράς ειδικά έκτακτα αλλά ο χρόνος και η εμπειρία μας δίδαξαν ότι στην πράξη πάντα χρειάζονται έκτακτα μέτρα στήριξης. Θα υπάρχουν τέτοιες συνθήκες ε, λόγω επιδημιών ε, των ζώων ή εμπορικών διαμαχών και απαιτείται η στήριξη στους αγρότες. Τώρα περνάμε στην τρίτη σύσταση το συνέδριο πρότεινε να φτιάξουμε μηχανισμούς και κριτήρια για να δούμε πότε θα πρέπει να εισαχθούν εξαιρετικά έκτακτα μέτρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει τονίσει και το Ελεκτικό Συνέδριο αλλά και διάφοροι πανεπιστημιακοί ότι πρέπει να έχουμε μέτρα τα οποία θα ε, έχουν έναν αυτοματισμό στις παρεμβάσεις αυτές. Ε, η Κομισιόν, ε, σε συμφωνία με Κοινοβουλή Κομισιόν, είπε ότι ποτέ θα φτάσουμε σε αυτή τη θέση, ποτέ δεν θα έχουμε μία συνταγή που θα καλύπτει όλες τις διάφορες συνθήκες για, που προκαλούν πτώση του εισοδήματος των αγορτών. Γι' αυτό ο κανονισμός της κοινή οργάνωσης αγοράς τα σχετικά άρθρα ε, προβλέπουν ε, μεγάλη ευελιξία. Αλλιώς ε, θα βρεθούμε χωρίς δυνατότητα παρέμβασης. Ή τα κριτήριά μας θα επηρεάζουν τη συμπεριφορά των αγορών. Αν υπήρχε ένα κριτήριο, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα προκαλούσε παρέμβαση, οι αγορές θα χειραγωγούσαν τις τιμές για να πετύχουν αυτόν τον στόχο και θα μας ανάγκαζαν να παρέμβουμε. Ε, δεν είμαστε υπέρ ε, μιας τέτοιας κατεύθυνσης. Παρόλα αυτά δεχόμαστε ότι το να έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια εξ άντε έχει κάποιους κινδύνους, αλλά παρόλα αυτά ε, πρέπει να το έχουμε κατά νου. Και τέλος για την τελευταία σύσταση για τα έκτακτα μέτρα στην ε, συγκεκριμένη περίπτωση αυτή και μιλάμε για μέτρα ε, που ελήφθησαν μετά το ρώσικο εμβάργο και στον τομέα των προκυπευτικών πράγματι τα έχουμε συζητήσει με το ελεκτικό συνεδρίο τη βάση δηλαδή της παρέμβασης και τις τιμές ε, απόστασης από την αγορά φρούτων και λαχανικών οπότε ουσιαστικά το θέμα αυτό το ήταν κάτω από τις τιμές της αγοράς και αν θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπεραντιστάθμιση. Όμως ε, είναι μια εξαιρετική περίπτωση, αλλά δεχόμαστε ότι πρέπει να το δούμε, <coughs> θα το επανεξετάσουμε στο πλαίσιο της δευτερογενούς ε, νομοθεσίας ε, που πρέπει να δημιουργηθεί για να αποφύγουμε το να προκύψουν ξανά τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον γιατί συμφωνούμε με το συνέδριο ότι ε, πρέπει να αποφευθεί η υπεραντισάθμιση όταν λαμβάνονται έκτακτα μέτρα. Βεβαίως, ε, συχνά σε καταστάσεις ανάγκης η προτεραιότητα είναι η ταχύτητα να δώσουμε το μήνυμα στις αγορές ε, της σταθερότητας και καμιά φορά γίνονται λάθη αλλά πρέπει να διδαχτούμε από αυτά τα λάθη. Αυτά κυρία Πρόεδρε και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι το ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστούμε πολύ την Κομισιόν. Ε, συνάδελφε Φλάνακαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Το να πω ότι έρχεται στο σωστό χρόνο ε, δεν αρκεί καν. Γιατί σήμερα το απόγευμα στις 2 θα έχουμε μια συνάντηση σκιωδών για την ΚΑΠ όπου θα συζητήσουμε ακριβώς αυτά τα άρθρα και προφανώς ε, θα συζητήσουμε το όφελος αυτών των μέτρων και με ποιον τρόπο θα πρέπει να εφαρμόζονται. Ένα από τα ερωτήματα που ανέκυψε και είναι αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ε, προήλθε από μια αριστερή πολιτική ομάδα, από εμένα, είναι αν θα πρέπει να βασίζονται οι απώλειες στον όγκο ή στην ε, αξία γιατί γενικά λιγότερο όγκο σημαίνει υψηλότερη τιμή. Και δεν έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένο συμπέρασμα τι θα, για το τι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ε, ενεργοποιούνται αυτά τα κονδύλια. Επίσης υπάρχει ε, μεγάλη ανησυχία από την κοινότητα των γεωργών σχετικά με το αν θα πρέπει να δίνονται άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς αν θα πρέπει να διπλασιάζονται από αυτό το καθεστώς και οι γεωργοί έχουν τους δικούς τους τρόπους μέσω των άμεσων ενισχύσεων για να μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις ε, από το τι μπορεί να τους φέρει το μέλλον. Υπάρχουν και διασυνδέσεις και με τραπεζικά ε, ιδρύματα κτλ. Προφανώς εσείς έχετε περιορισμένο, περιορισμένες δυνατότητες, αλλά εδώ επικεντρωνόμαστε στον κλάδο των οποροκυπευτικών ένας κλάδος ο οποίος ε, θα μπορούσε να είναι επικερδής. Θα ήταν ε, πολύ ενδιαφέρον να δούμε ε, αντίστοιχη έκθεση για τα γαλακτοκομικά και για το βόηο κρέας. Γιατί ειδικά σε αυτόν τον κλάδο πολλοί ε, δραστηριοποιούνται κάτω, με τιμές κάτω του κόστους. Θα μπορούσε κανείς να εικάσει γιατί το κάνει αυτό. Ένας από τους λόγους πάντως είναι ότι ο, η αγορά, για παράδειγμα, δεν, λαμβάζει, δεν λαμβάνει υπόψη τη αυτές τις υπηρεσίες. Οπότε οι ο υπολογισμός της αξίας στη βάση των τιμών της αγοράς είναι πολύ δύσκολος. Απλά αναρωτιέμαι πώς θα μπορούσε να αποφεληθεί ο κλάδος αυτός αν δεν υπάρχει, αν δεν προβλέπεται ε, και ένας κλάδος ε, κοινή ωφέλεια παραγωγής στην, στην ΚΑΠ. Εγώ λέω το εξή. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα, δεν θα μου δώσει λεφτά αν ε, βάλω εγώ φωτιά στο σπίτι μου. Αν, ε, κάτι αντίστοιχο όμω γίνεται με, με τα μέτρα αγορά. γιατί ακριβώς θα δημιουργηθούν προβλήματα για την ε, τιμή του βόηου κρέατος που παράγεται στην Ιρλανδία για παράδειγμα. Ήδη υπάρχει ένα ε, καθεστώς για το, ε, για το βόηο Αυτό ακολουθεί την ίδια ε, διαδρομή όπου δίνονται κίνητρα ε, στους γεωργούς στην Ιρλανδία ε, ύψους 50 εκατομμύριων ευρώ για την μείωση της παραγωγής τους. Το συνέδριο έχει άποψη για την αξιοπιστία των επιστημονικών δεδομένων της αποτελεσματικότητας ε, των κινήτρων αυτών για την μείωση της παραγωγής, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν. Και νομίζω ότι ο κύριος Σίνη είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον από την Κομισιόν και συμφωνώ μαζί του ότι είναι ανησυχητικά τα πράγματα γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου η αγορά θα χειραγωγεί την κατάσταση όπου θα ξεκινούν ε, εσφαλμένες, ψευδείς δηλαδή αιτήσει ασφάλισης. Και τέλος, Έχουμε ε, μια εξαιρετική συγκυρία αυτή τη στιγμή. Χθες στη ΣΥΠΑ έγινε μια συζήτηση για για την βιοποικιλότητα Ένα από αυτά που με ανησυχούν σχετικά αυτές τις ε, ασφάλειες για τη συγκομιδή είναι ότι τελικά καταλήγουν τα χρήματα αυτά σε διάφορους μεσάζοντες και εταιρείε. Τελικά μήπως αυτά τα χρήματα υπάρχει κίνδυνος να φτάσουν ε, σε τσέπες άλλων ανθρώπων πέραν από αυτούς για τους οποίους προορίζονται τα χρήματα αυτά. <laughs> Ναι, ήταν ε, μια θεμελιώδης ε, ανάλυση την οποία βεβαίως δεν θα μπορέσουμε να φωτίσουμε μόνο με τη βοήθεια αυτής της έκθεσης. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω αν και άλλα ε, μέλη της Επιτροπής μας έχουν σχόλια να κάνουν. Ο κύριος Αστέλ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική και να ευχαριστήσω και το ελεγκτικό συνέδριο για την ανάλυση και τον εισηγητή για την εισήγησή του, φυσικά την έκθεσή του και τις πρώτες απαντήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ελεκτικό συνέδριο συστήνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παρακινήσει τους γεωργούς να προετοιμάζονται καλύτερα, ε, να παρακολουθεί την ενίσχυση για την ασφάλιση, τα κριτήρια έναρξης και λήξης των εκτάκτων μέτρων, θα επανέλθω σε αυτό, και να προσαρμόσει τις αποζημιώσεις για τις ε, επιχειρήσεις απόσυρσης προϊόντων. Το συνέδριο θεωρεί ότι τα μέτρα τα οποία έχουν σκόπο να βοηθήσουν τους γεωργούς να προστατεύσουν ε, τα προϊόντα τους από τη μείωση τιμών και την απώλεια παραγωγής ε, δεν κατάφερε να επιτύχουν το στόχο τους και η χρήση τους είναι ισχνή και ε, άνηση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. μετά από τα πρώτα στοιχεία που μας απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπεύει να ξεκινήσει συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσει να ε, ε, διορθώσει αυτή την κατάσταση. Και κάποια στοιχεία για τα πάνω από 500 εκατομμύρια που δόθηκαν για τον τομέα των απορροκυπευτικών το διάστημα 2014-2018 σε απάντηση στο ρωσικό εμπάργο. Ήδη αναφέρθηκε το θέμα αυτό σήμερα το πρωί. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε καθορίσει κάποια κριτήρια και αντικειμενικές παραμέτρους για να δει κατά πόσον είναι εύστοχα τα μέτρα και αν θα πρέπει να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια αυτά. Σύμφωνα με το ελεγκτικό συνέδριο, το 61% της ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκε από τους παραγωγούς ε, μήλων, ενώ οι εξαγωγές μήλων ήταν μόνιμες ε, και μάλιστα ορισμένε φορές είχαμε και αύξηση. Ε, αυτό όμως δεν εμπόδισε τη διαδικασία να ολοκληρωθεί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόλις μας το είπε, θεωρεί ότι είναι μια έκτακτη περίπτωση Ακόμα βέβαια δεν έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα από αυτή την κακή διαχείριση του ρωσικού εμπάργου του 2014 και νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου στο μέλλον να μην έχουμε υπερβολικές αποζημιώσεις για τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λευτέρη, έχεις το λόγο. Να ευχαριστήσω και τον εισηγητή της έκθεσης, αλλά και το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πραγματικά αισθάνομαι ότι αγγίζουν το θέμα με ιδιαίτερη ευαισθησία, γιατί είναι γνωστό σε όλου μα ότι οι αγρότε είναι η, η ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, εκείνη η οποία συνεισφέρει σημαντικά στην ακαθάριστη χωρία παραγωγή. Είναι πολύ απαραίτητη η ύπαρξη των αγροτών και τη υπαίθρου, αλλά εν είναι ευάλωτη με αποτέλεσμα να αναζητούμε όλοι τρόπου σταθεροποίηση αυτού του εισοδήματο. Όμω πιστεύω ότι κάποιε απαντήσει δίνονται μέσα από τι ίδιε τι συστάσει του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου αλλά και τι διαπιστώσει. Δηλαδή, για μένα είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι αναφέρεται και γίνεται παραδεκτό από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο ότι τα, αυτά τα 41 δισεκατομμύρια που δίνονται για την κοινή γεωργική πολιτική δεν πάνε στοχευμένα σε αυτού που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δηλαδή, δεν δίνονται σε αυτού που έχουν την ανάγκη για να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν καλύτερα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαπίστωση που πρέπει να υπάρξει και περαιτέρω ανάλυση, αλλά πολύ σημαντικό να εξευρεθεί και τρόπο αποτελεσματικό για να πηγαίνουν στοχευμένα τα χρήματα σε αυτού που πραγματικά έχουν ανάγκη για να μπορέσουν να αναπτυξούν και να αναπτύξουν και το γεωργικό τομέα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι η αναποτελεσματικότητα που υπήρξε εξαιτία πιθανώ και τη αδυναμία των κινήτρων να υπάρξει σύνδεση των γεωργών με το περιβάλλον. Δηλαδή, μέσα στα πλαίσια μια ευρεία προσπάθεια που γίνεται για αναχέτηση τη κλιματική αλλαγή, οι γεωργοί πρέπει να αποτελέσουν μέρο αυτή τη προσπάθεια και το ότι μέχρι σήμερα φαίνεται ότι δεν έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και ένα τρίτο που θέλω να, έτσι να αναφέρω είναι ότι η αναποτελεσματικότητα στο να υπάρξει η ασφάλιση των γεωργών μα, αφού απέτυχε σε 17 κράτη-μέλη και μόνο το 8% των αγροτών στηρίζονται από την ευρωπαϊκή ασφάλιση, με ποιο τρόπο αυτό θα γενικευθεί και με ποιο τρόπο πραγματικά θα δοθεί απάντηση στο σημαντικό ερώτημα που τίθεται μέσα από την έκθεση για σταθεροποίηση του εισοδήματο των αγροτών μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλες παρεμβάσει. Όχι προς το παρόν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο ξανά στο ελεγκτικό συνέδριο για να απαντήσει στα όσα υπόθηκαν από τους συναδέλφους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να απαντήσω στα ερωτήματα που έθεσε και ο κύριος Φλάναγκαν. Αν κατάλαβα σωστά, το πρώτο ερώτημα ήταν αν, αν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τον όγκο ή την αξία όταν λαμβάνονται έκτατα μέτρα. Αυτό εξαρτάται από το στόχο του μέτρου. Αν ο στόχος είναι το εισόδημα, τότε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα δύο. Αν, υπάρχουν, αν υπάρχει κάποιο άλλο στόχο, μπορεί να γίνει μια συζήτηση διαφορετικά. Για, τα, για τον κλάδο των γαλακτοκομικών και του βόηου κρέατο, εμεί αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν έλεγχο για τα γαλακτοκομικά ε, θα έχουμε μια σχετική ειδική έκθεση σε λίγους μήνες. Για το βόλιο κρέας δεν έχει ξεκινήσει κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια καλή ιδέα. Όσον αφορά την, ε, τις επιστημονικές ενδείξεις για τη μείωση τη παραγωγής, εγώ δεν μπορώ να σας δώσω ε, στοιχεία για το βόλιο κρέας, γιατί δεν έχουμε κάνει έλεγχο. Όμω, μπορώ να σας υπενθυμίσω αυτό που λέμε στην έκθεση μα όσον αφορά τα απορροκυπευτικά, και την αποζημίωση για τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Στην Ισπανία και η Ελλάδα αποζημιώθηκαν για την παραγωγή ε, νεκταρινιών, ροδακίνων και ταυτόχρονα η Ιταλία προσπαθούσε να μειώσει την παραγωγή αυτών των συγκεκριμένων φρούτων. Οπότε θέτουμε και ορισμένα ε, ερωτήματα σχετικά με το αν υπήρξε σωστός συντονισμός κάποιο να αποζημιώνεται και κάποιο άλλο να, να. ενώ υπάρχει μια προσπάθεια να μειωθεί η παραγωγή, παρόλα αυτά να δίνονται και αποζημιώσει. Για την ασφάλιση, εγώ θα ήθελα να αναδείξω τρία θέματα. Έχουμε μια περίπτωση στην έκθεσή μας από τις ΗΠΑ όπου οι αγρότες ασφαλίζονται παράγουν τις οδιές τους με λιγότερο ανθεκτικό τρόπο από εκείνους που δεν είναι ασφαλισμένοι. Γιατί ξέρουν ότι ό,τι και να συμβεί θα πάρουν αποζημίωση από την ασφάλιση. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Η ασφάλιση θα πρέπει να συνάπτεται με, ταυτόχρονα με τους όρους που θα εξασφαλίζουν ότι οι αγρότες θα παίρνουν κάποια προληπτικά μέτρα. Όπως είναι η εναλλαγή των καλλιεργιών, για παράδειγμα, που θα μπορούσε να, να εξασφαλίσει ότι πραγματικά θα ωφεληθούν από την, από την παραγωγή τους και όχι να βασίζονται στην αποζημίωση. Τρίτο στοιχείο όσον αφορά τις ε, ε ασφαλίσεις είναι δεδομένου και κιόλας ότι τα κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις όπως φαίνεται και στο χάρτη. Υπάρχουν και χώρες που δεν ε, βασίζονται σε ευρωπαϊκά κονδύλια για την ασφάλιση. ασφάλιση. Κάποια κράτη-μέλη έχουν και εθνικά συστήματα. Κάποια άλλη ε, δεν δίνουν καθόλου στήριξη γιατί η, η, ε, η αγορά εξασφαλίζει την ασφάλιση αυτή. Γι' αυτό Γι' αυτό και εμεί ε, κάνουμε σύσταση προ την Κομισιόν ότι δεν υπάρχει στοιχείο, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι θα υπάρχει ε, ότι υπάρχουν ωφέλη από την χρήση ενωσιακών ε, κονδυλίων για την παροχή αυτής της ασφάλισης, αφού αυτή μπορεί να παρέχεται από την, από την αγορά. Αυτό προτείνουμε και προς την Κομισιόν. Στο μέλλον με την κλιματική αλλαγή τίθεται και το ερώτημα αν όλο και περισσότεροι αγρότες θα πληγούν από ξηρασίες, πλημμύρες κτλ. Γιατί σε αυτή την περίπτωση προφανώς η ασφάλιση θα γίνει πιο ακριβή. Και το ερώτημα είναι πότε, που, πότε ακριβώς θα ε, συναντήσουμε το σημείο καμπής ε, εκεί που η ασφάλιση πια δεν θα μπορεί να καλύψει τις απώλειες. Γι' αυτό και χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στην, ε, στην, στα προληπτικά μέτρα ώστε να, τα προληπτικά μέτρα να είναι πιο ισχυρά από την ασφάλιση. Συμφωνούμε πάντως με την Κομισιόν ότι τα καθεστώτα ενίσχυσης είναι το βασικό έργαλο, εργαλείο για να εξασφαλιστεί η επιβίωση των αγροτών ακόμα και σε ακραίες καιρικέ συνθήκες. Να ευχαριστήσω και εγώ την Κομισιόν για όλες τις επαφές που είχαμε στις συναντήσεις μας, στη διάρκεια των ελέγχων Συζητήσαμε αυτά τα θέμα διεξοδικά. Εντάξει, σε κάποιες συστάσεις καταλήγουμε ενδεχομένως σε ελαφρώς διαφορετικές στάσεις, ε, θέσεις. Ε, είναι ευθύνη της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου τώρα να καθορίσουν τι ακριβώς θα γίνει. Κάποια κράτη-μέλη ήδη έχουν ε, αρχίσει την εφαρμογή των συστάσεων μας. Η Γαλλία και η Ιταλία, για παράδειγμα, έχουν καταρτήσει σαφείς προϋποθέσεις για το πότε εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα Οπότε δεν θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και όσον αφορά τις τιμές της αγοράς, αυτές είναι πάντοτε γνωστές, οπότε ε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει πρόβλημα να ε, εισαγάγει κανείς τέτοια μέτρα. Δεν ξέρω αν, ε, από τον κύριο Σαντέλη και τον κύριο Χριστοφόρου υπήρξαν κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα προς εμάς. Δεν μπόρεσα να παρατηρήσω κάτι τέτοιο. Αν ξεχνώ κάτι παρακαλώ πείτε το μου και θα σας απαντήσω ευθύ αμέσως. Ωραία. Να ρωτήσω τους συναδέλφους αν υπάρχουν ερωτήσεις προς το Ελληνικό Συνέδριο και προς την Κομισιόν. Ο συνάδελφος Φλάναγκαν. Όχι. Νομίζω ότι ήταν πλήρες όπως πάντα. Ε, έχω πολλά πράγματα να επικρίνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε γενικές ε, γραμμές πρέπει να πω ότι με εντυπωσιάζει το ελεγκτικό συνέδριο. Η Κομισιόν θέλει να πει κάτι άλλο. Ο κύριο Κανέλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάποιε γενικέ παρατηρήσεις. Ανέφερα προηγουμένως ότι θα πρέπει να αποφύγουμε να δημιουργήσουμε την εντύπωση ότι η λύση ίσως ε, στο να παρέχουμε στήριξη στους γεωργούς και να αποφύγουμε πιθανές ε, διαταραχές ε, είναι να έχουν όλοι ασφαλιστική κάλυψη αυτό ποτέ δεν θα είναι η λύση και νομίζω ότι ο κύριος Φλάναγκαν εξήγησε και την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες που γίνεται πιο εκτεταμένη η χρήση ασφάλισης και δεν νομίζω ότι το λέγατε ως κάτι θετικό, αλλά για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο τομέας των ασφαλιών των Ηνωμένων Πολιτειών παίρνει το 15% της στήριξης για την ασφάλιση των ε, ε εσοδιών ως ε, ίδιο εισόδημα. Ουσιαστικά δεν παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη δωρεάν. Αν λοιπόν ακολουθήσουμε και εμεί αυτό το μοντέλο, και έχουμε ένα μόνιμο πόρο, ε, ουσιαστικά ένα τμήμα αυτών των χρημάτων θα περάσει στον ασφαλιστικό κλάδο. Πολύ ευχαρίστω βεβαίω θα το λάβουν, αλλά θα προτιμήσουμε θα, να δοθεί στου γεωργού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν στηρίζουμε και την περίπτωση ε, αν οι γεωργοί θέλουν να έχουν κάποια ασφαλιστική κάλυψη ή να καλύπτουν και κάποια αμοιβαία κεφάλαια. Γι' αυτό και στι προτάσει, στον πυλώνα 2, είναι υποχρεωτικό για τα κράτη-μέλη να προβλέψουν τουλάχιστον για τους γεωργούς και τις οργανώσεις παραγωγών κυρίως τη δυνατότητα να ε, έχουν ε, τέτοια κάλυψη. Και ιδιαίτερα τα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία διαφέρουν από την ασφάλιση, ε, παρέχουν μια σειρά από ενδιαφέρουσες επιλογές που έχουν χρησιμοποιηθεί με κάποια επιτυχία, ιδιαίτερα στη Γαλλία και στην Ιταλία, Εκεί οι γεωργοί και οι οργανώσεις παραγωγών είναι οι ίδιοι αρμόδιοι, τα διαχειρίζονται μόνοι τους και ιδιαίτερα στον τομέα των απορροκυπευτικών, αλλά όχι μόνον, είναι ένα αποτελεσματικός τρόπος να αποφεύγουν ε, προβλήματα από τον καιρό, από ε, ζυζάνια ή και τις ίδιες τις διακοιμάνσεις της αγοράς. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πολύ ευχαρίστω θα θέλαμε να στηρίξουμε και θα θέλαμε να επεκταθεί. Και τέλος, όσον αφορά τις υπερβολικές ε, αποζημιώσεις, το ελεγκτικό συνέδριο Δικαστήριο έκανε πολύ ε, σημαντικέ συστάσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ναι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ε, ε, στα έκτακτα μέτρα στήριξη υπάρχει ο κίνδυνο και σε κάποιε περιπτώσει μπορεί να υπερβήκαμε και τα όρια. Ειλικρινά είναι δύσκολο να το αποφύγει κανείς αυτό όταν παρεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσης. Για το παράδειγμα της Ρωσίας, να μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι επέβαλαν εμπάργο στις ευρωπαϊκές εξαγωγές αν συνέπειες για 5 δις ευρώ εμπορίου. Ήταν σκεμμένη επιλογή για να κάνουν τη μέγιστη δυνατή ζημιά στον τομέα των εξαγωγών των γεωργικών και διατροφικών προϊόντων και δεν μπορούσε να αδρανίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην παρέμβει. Γι' αυτό και κάναμε ό,τι κάναμε. Και νομίζω ότι ε, μακράν στον τομέα των ε, ε, ζωικών προϊόντων νομίζω ότι η παρέμβαση ήταν επιτυχής. Αναγνωρίζουμε ότι στον τομέα των απορροκυπευτικών ήταν λίγο πιο πιο θολά τα πράγματα, αλλά μαθαίνουμε και εμείς από την εμπειρία και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου φυσικά είναι τμήμα όλης αυτής της διαδικασίας μάθησης και θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. So, ein ganz herzliches Dankeschön. Ευχαριστώ λοιπόν ε, πάρα πολύ και τώρα κανονικά πρέπει να συζητήσουμε το επόμενο θέμα αλλά λείπει το μέλος του ελεκτικού συνεδρίου οπότε κάνουμε διάλειμμα 10 λεπτών. 5 λεπτών. Λοιπόν, 5 λεπτά μέχρι να έρθει. As he just arrived. <laughs> We are a little bit quicker than foreseen in the agenda, so... Λοιπόν, ε, το είχαμε προβλέψει στην ημερήσια διάταξη και ήταν κάπως δύσκολο. Καλό, guten Morgen. Ναι, καλημέρα σας. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίζω το μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, τον κύριο Τάκουλα. Ε, βιαστήκαμε σήμερα, πήγαμε πιο γρήγορα και σας δυσκολέψαμε. Διότι ε, ξεκινήσαμε ήδη με το σημείο 6 την ε, έκθεσή σας 25.019 ε, ποιότητα των δεδομένων στο πλαίσιο της δημοσιονομικής στήριξης αδυναμία σε ορισμένους δείκτες και επαλήθευση των πληρωμών μεταβλητών δόσεων. Η συγητή είναι ο κύριος Χριστοφόρου. Θα σας ε, δώσω το λόγο λοιπόν. Thank you, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερος ε, που είμαι πάλι στην ε, Επιτροπή μας. Είχα έρθει τελευταία φορά εδώ ως βουλευτής, αλλά τώρα είμαι με ένα νέο ρόλο. Θα σας μιλήσω για την ποιότητα των δεδομένων. Θα δούμε λοιπόν αν η Κομισιόν βασιζόταν ε, σε αξιόπιστα δεδομένα όταν έδινε δημοσιονομική στήριξη. Εξετάσαμε 24 τέτοιες συμβάσεις σε 8 χώρες με τις μεγαλύτερες πληρωμές το 2017. Οι 24 αυτές συμβάσεις περιλάμβαναν οι 248 δείκτες απόδοσης από αυτές τις 8 χώρες. Έγιναν επιτόπιες επισκέψεις σε 3 την ε, Ιορδανία, τη Γεωργία και την Βολιβία. Όπως βλέπετε από τον τίτλο της έκθεσης, ήταν ε, τεχνικός ο έλεγχος, ε, αφορούσε την αξιοπιστία και ακρίβεια των δεδομένων από διάφορα έγγραφα. Δεν αξιολογήσαμε το εάν η στήριξη του προπολογισμού στήριξε αποτελεσματικά τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές. Ποια ήταν λοιπόν τα κύρια ευρήματα. Εν ολίγης, ε, οι δείκτες λειτουργούν και η επαλήθευση το ίδιο. Πρώτα θα αναφερθώ στους δείκτες και μετά στην επαλήθευση της Κομισιόν. Όσον αφορά τους δείκτες, το πρώτο θετικό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι οι δείκτες ήταν ευθυγραμμισμένοι με τις στρατηγικές των χωρών και τις αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά δυστυχώς 87% αυτών ήταν ε, δείκτες εργασιών ε, ή αποτελέσματος ε, και μόνο 13% αφορούσαν το αποτέλεσμα ή τον αντίκτυπο, δηλαδή μακροπρόθεσμοι δείκτες. Επιπλέον, πρέπει να είναι συγκεκριμένοι οι δείκτες να έχουν μετρήσιμους στόχους και όταν αυτό γίνεται να έχουν και ένα αξιόπιστο σημείο αναφοράς ως αφετηρία. Αλλιώς δεν μπορούμε αντικειμενικά να μετρήσουμε την πρόοδο που κάνουν οι χώρες αυτές πριν ε, ε, πληρώσουμε μεταβλητές δόσεις. Είδαμε ότι ένα τρίτο των δικτών δεν επέτρεπαν αντικειμενική μέτρηση των ε, αποτελεσμάτων. Παραδείγματο χάρη, 29% των δικτών δεν ήταν αρκετά συγκεκριμένοι. Χρησιμοποιούσαν παραδείγματο χάρη γενικολογίε όπως να βελτιωθεί ή να αυξηθεί η έμφαση. Επίσης Επίση υπηρχε πρόβλημα με, το με τη βάση αναφοράς. Ε, π.χ. μιλούσε για μία 10% ε, αύξηση, ξέρω εγώ, σε όσους έλαβαν στήριξη. Βρήκαμε το 41% των περιπτώσεων η αφετηρία ε, είτε δεν υπήρχε είτε δεν ήταν επαρκής. Επίσης. το θέμα ήταν το εάν ε, υπήρχαν τα απαραίτητα κίνητρα για να γίνουν οι κατάλληλες μεταρρυθμίσεις. Οι περισσότεροι δείκτες ε, είχαν σωστή ισορροπία μεταξύ του να είναι φιλόδοξοι και εφικτοί και είχαν το κατάλληλο αποτέλεσμα. Υπήρχαν κάποια παραδείγματα όπου οι στόχοι ήταν πολύ εύκολοι ή χρησιμοποιούσαν λάθος σημεία αφετηρίας. Βρήκαμε ακόμα και μια περίπτωση στη Ρουάντα όπου η πρόταση περί ηλεκτρισμού από ΑΠΕ είχε ως αποτέλεσμα μείωση της σχετικής παραγωγής, αλλά η Κομισιόν παρόλα αυτά πλήρωσε. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω κάποια ευρήματα για το δεύτερο τμήμα του ελέγχου μας, ε, την επαλήθευση δηλαδή που κάνει η Κομισιόν όταν πληρώνει μεταβλητές δόσεις. Η ευθυρία των πληρωμών είναι ένα αίτημα από τις ε, χώρες αυτές, βασίζεται στα δεδομένα ιδίων των χωρών. Οπότε τα συστήματα αυτά είναι οι πατογενείς πηγές πληροφοριών για την απόφαση πληρωμών. Και δεν προξενεί εντύπωση ότι κάθε χώρα έχει τη δικιά της μέθοδο για την συλλογή, ανάλυση και χρήση δεδομένων και τις ε, δικές της δυνατότητες. Συνεπώς, ε, πριν ξεκινήσουμε τις ε, σχετικές επιχειρήσεις, η Κομισιόν πρέπει να αξιολογήσει το σύστημα το οποίο υπάρχει για την κατάρτιση δικτών που αργότερα θα χρησιμοποιηθούν για τέτοιες ε, πληρωμές. Βρήκαμε ότι η αξιολόγηση της Κομισιόν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση συστημάτων πράγματι αξιολόγησε τα απαιτούμενα στοιχεία, αλλά η Κομισιόν Παριτά συμπεραίνει κάποια πράγματα για την αξιοπιστία των ε, δεδομένων η οποία δεν είναι ικανοποιητική. Όσον αφορά την επαλήθευση της αξιοπιστίας των δεδομένων, το γενικό μας συμπέρασμα ήταν ότι η Κομισιόν δεν έκανε πάντα επαλήθευση Ε, είδαμε ότι ε, κάποιες διαδικασίες επαληθευσής δεν ήταν σωστές, δεν υπήρχε η κατάλληλη ε, βεβαιότητα για να προχωρήσουν στις πληρωμές. Σε έξι συμβάσεις από τις 24 ελήφθη το αίτημα μαζί με τα δικαιολογητικά αλλά η Κομισιόν δεν έκανε αποτελεσματική επαλήθευση των σχετικών δεδομένων για την πληρωμή. Αυτό έγινε κυρίως επειδή η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασιζόταν στην ακρίβεια των δεδομένων που έδιναν οι χώρες εταίροι ή στην επαλήθευση που έκαναν εξωτερικοί ειδικοί ε, για λογαριασμό της Κομισιόν χωρίς οποιαδήποτε επαλήθευση των δεδομένων από την ίδια την Κομισιόν. Από συνολικά 234 εκατομμύρια ευρώ πληρωμών μεταβλητών δόσεων συμπεράναμε ότι τα δεδομένα που έδιναν οι χώρες εταίροι δεν δικαιολογούσαν την επίτευξη των ε, δικτών για την πληρωμή 13,3 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον είδαμε ότι η Κομισιόν πλήρωσε 3,4 εκατομμύρια σε δύο χώρες με βάση δείκτες που είχαν λάθος σημεία αφετηρίας. Παρά το ότι υπήρχε συμβατική υποχρέωση ε, να πληρωθούν καθώς είχαν επιτύχει τον στόχο δεν είχε επιτευχθεί καμία πραγματική πρόοδος. Κυρία Πρόεδρε, συνοψίζοντας, καταλήξαμε ότι για το 1 τρίτο των δικτών η σημασία τους ε, υπονομευόταν από την διατύπωση και δεν μπορούσε να μετρηθεί αντικειμενικά το αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση της Κομισιόν για το εάν είχαν ε, επιτευχθεί οι δείκτες για τις μεταβλητές δόσεις δεν ήταν πάντα αξιόπιστη. Θα ήθελα λοιπόν καταλήγοντας να ευχαριστήσω την Κομισιόν καθώς δέχτηκε όλες τις συστάσεις μας και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάκουλα. Ο κύριος Χριστοφόρου είναι ο εισηγητής. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θέλετε να μιλήσετε τώρα ή να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτιμάτε να μιλήσουμε με την Κομισιόν πρώτα. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση να δώσω το λόγο στην κυρία Νάταλη Μπραχάρ εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε τον λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι προβουλευτές, μέλη της, του Ελληνικού Συνεδρίου. Τα συστήματα δημοσιονομικής στήριξης ε, κατευθύνονται προς την ανθεκτικότητα, όπως λέει και το συνέδριο. Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν συνεργάζεται στενά με χώρες εταίρους για να προσδιορίζει τομείς ε, και δείκτες που προκύπτουν από τους ίδιους τους κλάδους μέσω του στρατηγικού πλαισίου που έχει συναυθεί με την χώρα εταίρο για τον καθορισμό αξιόπιστων ε, ε, στόχων με την συλλογή αξιόπιστων δεδομένων από την χώρα. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσεκτικός προγραμματισμός, σχεδιασμός και συνεχής παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών. Γι' αυτό τον λόγο η Κομισιόν χαιρετίζει την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που καταρτίστηκε με πολύ επικοδομητικό τρόπο και επικοδομητικό πνεύμα. Η Κομισιόν αποδέχεται όλες τις συστάσεις οι οποίες θα είναι χρήσιμες στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων δημοσιονομικής στήριξης Και αυτό είναι ε, κάτι το οποίο το, ε, το υπηρετούμε ως στόχο εδώ και πολλά χρόνια. Η στάση της Κομισιόν απέναντι στις στρατηγικές με τις χώρες εταίρους ε, είναι συνεπής, που δείχνει σαφή κατεύθυνση προς την επίτευξη αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων. Στο πνεύμα αυτό καθορίζουμε στόχους με τις ε, ε, χώρες εταίρους που προκύπτουν συνήθως από τη στρατηγική των ίδιων των χωρών και μια από, ε, ένας από τους βασικούς στόχους της δημοσιονομικής στήριξης είναι η ενίσχυση των συστημάτων και των θεσμικών ικανοτήτων των χωρών εταίρων συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που έχουμε για την δυνατότητα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, πολλοί από τους δείκτες της Κομισιόν ενισχύουν αυτούς τους ε, στόχους και η έκθεση αυτή είναι ε, ισορροπημένη περιγράφοντας τι πρέπει να γίνει στο μέλλον συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων που χρειάζονται ε, σε ορισμένες περιπτώσεις για τους δείκτες και τους στόχους αφετηρίας. Κομισιόν ήδη εργάζεται για την βελτίωση της στήριξης που παρέχεται σε χώρες εταίρους όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και την βελτίωση των ε, στατιστικών και διοικητικών δεδομένων τους. Θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη διασφάλιση ποιότητας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ε, δείκτες για την ποιότητα θα διατυπώνονται με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων και των ε, ε, σημείων αφετηρίας. Και θα ενισχυθεί η συνολική ε, συνεργασία μας με τις χώρες εταίρους για την βελτίωση της αξιοπιστίας των δεδομένων. Περαιτέρω, για την βιωσιμότητα της στήριξής μας είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι ικανότητες των χωρών εταίρων για την παραγωγή ε, μετρήσιμων και συγκρίσιμων στοιχείων, όχι μόνο για τη δημοσιονομική στήριξη, αλλά και για την παρακολούθηση της εφαρμογής ε, των ε, δημόσιων πολιτικών. Συνολικά λοιπόν η Κομισιόν αναγνωρίζει τον, την επικοδομητική στάση που επιδεικνύει το ελεγκτικό συνέδριο κατά τη διάρκεια του ελέγχου που διενήργησε και χαιρετίζουμε τις συστάσεις για τη βελτίωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων και για την ενίσχυση της ικανότητας των χωρών εταίρων για την παραγωγή στατιστικών και διοικητικών δεδομένων. Τέλος, θα ήθελα να υπενθυμίσω δύο πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης. Πρώτον, είναι η συνέχεια που δόθηκε στην ειδική έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου 35 του 2016 σχετικά με τη χρήση της δημοσιονομικής στήριξης για την ε, βελτίωση της ε, ε, εγχώριας δημοσιονομικής ικανότητας στην υποσαχάρια Αφρική. Υπενθυμίζουμε ότι η Κομισιόν έχει λάβει όλα τα μέτρα που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο δράσης της Αντίσα Μπέμπα στο πλαίσιο συνεργασίας, ιδίως στα προγράμματα δημοσιονομικής στήριξης. Δεύτερον είναι η νέα έκθεση 19 για τη δημοσιονομική ε, στήριξη που πρόσφατα παρουσιάστηκε στις 3 ε, Δεκεμβρίου στην Επιτροπή ΔΕΒΕ όπου παρέστησαν ε, και οι Επιτροπές ΑΦΕΤ και ΚΟΝΤ. Και τα αποτελέσματα αυτής της ειδική έκθεσης είναι πολύ θετικά και δείχνουν την ανάγκη να συνεχιστεί η δημοσιονομική στήριξη ε, στην κατεύθυνση της ε, επίτευξης των στόχων για την βιώσιμη ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε τώρα στον εισηγητή. Κύριε Χριστοφόρου, έχετε το λόγο. Ε, καταρχήν θα εκφράσω την ικανοποίησή μου για τον θετικό τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει και τις εισηγήσεις και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου αυτό αποδεικνύει όχι μόνο το στοιχείο της συνεργασίας, αλλά και την ε, πρόθεση όλων να αντιμετωπιστούν θετικά εκεί και όπου υπάρχουν ελλείψεις, κενά, λάθη, παραλήψεις, ιδιαίτερα όταν αυτές οι επισημάσεις ε, ε, έρχονται από το ελεκτικό, Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Ταυτόχρονα να ευχαριστήσω για την εξαίρετη πραγματικά προσέγγιση και εκπόνηση αυτή τη έκθεση από το μέλο του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, του κ. Χάνου Τακούλα, και ιδιαίτερα δε για τις ξεκάθαρες επισημάσεις του. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι κάθε χρόνο προσφέρει 1,7 δισεκατομμύρια για χώρες μέλη εταίρους, τα οποία φαίνεται ότι αυτές οι μεταβλητές δόσεις είναι απαραίτητες γιατί αποτελούν το κίνητρο για την πρόοδο και στην υλοποίηση της ανάπτυξης αυτών των χωρών μελών. Όμως πρέπει να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με όσα οικονομικά προβλήματα και δυσκολίες έχει, και που ουσιαστικά αυτά είναι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών, ε, καθίσταται ο πρώτος στην παγκόσμια κλίμακα χορηγός δημοσιονομικής στήριξης σε χώρες μέλη. Άρα αυτά τα χρήματα για μας είναι ιερά και πρέπει να παρέχονται με φιδόν, με αποτελεσματικότητα, με αντικειμενικότητα, με ακρίβεια και να μην επιτρέπεται καμία διασπάθηση και καμία κακή διαχείριση από χώρες μέλη. Θεωρώ ότι χώρες, ε, από χώρε εταίρου. Χώρε οι οποίοι για οποιουσδήποτε λόγου δεν αξιοποιούν σωστά αυτά τα χρήματα ή καθίστανται προϊόν διαφθορά ή και εξαπάτηση, πρέπει να αποκλείονται εξ από το πρόγραμμα. Πολύ ορθά επισημάνθηκε, και αυτό είναι και ανησυχητικό, ότι σε τεχνικό επίπεδο το 1 τρίτο των διχτών ε, δεν εξασφαλίζουν αντικειμενικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Μάλιστα, πολύ εύστοχα, ο εισηγητή εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, και τον συγχαίρω γι' αυτό, αναφέρει ότι οι ελεκτέ διαπίστωσαν επίση ότι στι περισσότερε περιπτώσει η Επιτροπή δεν εξήγαγε ρητά συμπεράσματα σχετικά με την ικανότητα των χωρών εταίρων να παράγουν ακριβή δεδομένα. Τα κύρια ζητήματα στα οποία επικεντρώνονται αφορούν την εκπρόθεσμη επίδευση των τιμών στόχου, αποτελέσματα που μετρούνται βάσει εσφαρμένων τιμών βάση εσφαρμένη ελλειπή αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των δικτών, καθώ και τιμέ στόχου που δεν επιτεύχθηκαν καθόλου. Αυτό για μένα είναι εξόχω ανησυχητικό. Όπω ανησυχητικό είναι το ότι υπάρχει ομολογία ότι το 1 τρίτο των δικτών δεν εξασφαλίζουν αντικειμενικά μετρήσιμα αποτελέσματα. Δείχτε που είναι ανεπαρκεί και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν αντικειμενικά αποτελέσματα ή πρέπει να καταργούνται ή πρέπει να βελτιώνονται άμεσα. Είναι αδιανόητο το 87% των δικτών, όπω ελέγχθηκε, να είναι δείχτε διαδικασίες και να είναι μόνο το 13% δείχτε που προνοούν τα αποτελέσματα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφενός με για να διαφυλαχθεί αυτό το πρόγραμμα για τι μεταβλητέ δόσεις που είναι σημαντικές για τι χώρους εταίρου, για να διασφαλίσουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογούμενων πολιτών πάνε σε σωστό και στοχευμένων τρόπων και αξιοποιούνται αποτελεσματικά από χώρε που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Είναι χώρε που έχουν ανάγκη και το τελευταίο ευρώ. Άρα θεωρώ κομβική επισήμαση του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, όπου αναφέρεται ότι προτού εκταμιευθεί οποιοδήποτε ποσό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μεριμνά περισσότερο, ούτω ώστε να έχει στη διάθεσή τη τα σωστά δεδομένα. Ανησυχώ γιατί ουσιαστικά είναι σαν να εκφράζεται ότι γίνονται εκταμιεύσει χωρίς να υπάρχουν αυτά τα σωστά δεδομένα πριν να γίνει αυτή η εκταμίευση. Για μένα είναι κανόνας και όρο απαράβατος για την προστασία του ευρωπαϊκού χρήματος οπωσδήποτε να γίνεται διπλός και πολλαπλός έλεγχος πριν να εκταμιευθεί έστω και ένα ευρώ. Ταυτόχρονα θα θέσω ακόμα μια άλλη διάσταση που δεν ξέρω πόσο συνάδει, αλλά θα τη θέσω για να επιλεχθούν αυτές οι χώρες εταίροι και να τους δίνονται τα χρήματα. Γίνονται επισημάσεις και όσον αφορά το κράτος δικαίου που εφαρμόζεται σε αυτές τις χώρες, η δημοκρατία, η ισότητα αντρών γυναικών, ο σεβασμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή, γίνονται, ή δίνονται χωρίς να υπάρχει αυτός που για μένα έπρεπε να είναι ένας βασικός δείχτης. Παρά τα αυτά, κλείνοντας θέλω να επισημάνω ότι πράγματι γίνεται εξαιρετική δουλειά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, όμως μπορεί να βελτιωθεί όλη αυτή η εργασία εάν υιοθετηθούν οι επισημάσει του αγαπητού μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου του κ. Τακούλα και χαίρομαι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αποδέχεται εκ των προτέρων, ευερπιστώντα ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χριστοφόρου. Δεν ξέρω αν ο κύριος Στάκουλα θέλει να σχολιάσει κάτι. Παρακαλώ. Sí, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι πραγματικά μου άρεσαν αυτά που είπε ο κύριος Χριστοφόρου. Είμαστε νομίζω στην ίδια οπτική γωνία και είναι πολύ σημαντικό να το διαπιστώνει κανείς αυτό. Νομίζω ότι η βάση αυτού του ελέγχου είναι ότι αν χρησιμοποιείται στήριξη από τον προϋπολογισμό, υπάρχουν δύο πράγματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, κατάλληλοι δείκτες και δεύτερον, κατάλληλοι έλεγχοι πριν ε, γίνουν οι ε, πληρωμές ε, από τη στήριξη του προπολογισμού. Και ακριβώς αυτό επεσήμανε και ο εισηγητής, ο κύριος Χριστοφόρου. Και νομίζω ότι αυτό που θα ήθελα να πάω και επισημαίνω είναι ότι είμαι πολύ ικανοποιημένο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη και δέχεται όλες μας τις συστάσεις και ελπίζω στο μέλλον όταν και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη στήριξη του προπολογισμού ως ε, και πηξίδα ε, να γίνονται σωστά ε, όλα αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Η δημοσιονομική στήριξη ήταν πάντοτε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα και χάρη στο ελεγκτικό συνέδριο ε, νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά βελτιωτικά βήματα ακόμη και αν δεν είναι τέλεια τα πράγματα ακόμη. Στόχος είναι πάντοτε τα χρήματα να κατευθύνονται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Εμείς θα συνεχίσουμε βεβαίως ε, να παρακολουθούμε το θέμα, γιατί ιδίω ε, σε σχέση με τρίτες χώρες είναι πάντοτε περίπλοκο και δύσκολο και να δίνεις χρήματα και να παρακολουθείς το τι τελικά έγιναν αυτά τα χρήματα, που αξιοποιήθηκαν δεδομένου και ότι δεν έχουν πάντοτε όλες οι χώρες ακριβώς την ίδια αντίληψη με μας για το τι είναι η δημοκρατία, η νομιμότητα, η κοινωνική ε, οργάνωση. Ε, οπότε από αυτή την άποψη σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συστάσεις σας και για την αξιολόγηση στην οποία ε, καταλήξατε. Θα κάνουμε ένα τρίλεπτο διαλυματάκι τώρα, γιατί είχαμε πίσω στους συναδέλφους του επόμενου θέματος ότι θα το συζητήσουμε στις 11, θέμα σχετικά με την εικαζόμενη απάτη, ε, κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω οργανωμένου εγκλήματος στην Ιταλία. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε νωρίτερα από ότι είχαμε ε, πει στους συναδέλφους ότι θα ξεκινήσουμε. Ας κάνουμε ένα πεντάλεπτο διαλυματάκι, ίσως μπορούμε να πιούμε και ένα σύντομο καφεδάκι και 11 και κάτι ξεκινάμε. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Συνάδελφοι, να σας ε, παρακαλέσω είτε να μείνετε εδώ στην αίθουσα είτε να αποχωρήσετε ό,τι θέλετε. Περνάμε στο επόμενο σημείο της σα διάταξης το υπαριθμόν 7, συνέχεια που δόθηκε σε πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με εικαζόμενη απάτη στον τομέα των γεωργικών χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιταλία. Πολλά ΜΜΕ αναφέρουν, σήμερα μάλιστα και το πολίτικο, σχετικά με απάτες που σχετίζονται με τη μαφία στον γεωργιακό τομέα που έχει οδηγήσει και σε συλλήψει στην Ιταλία. Έχουμε λοιπόν σήμερα μια ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής και της Όλαφ και θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις υποθέσεις αυτές. Εγώ διάβασα το άρθρο στο Πολίτικο και πραγματικά αν το διαβάσει κανείς ε, φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σοβαρή η υπόθεση αυτή γιατί το οργανωμένο έγκλημα φαίνεται να ασκεί πίεση σε απλούς πολίτες για να μπορούν να, να μην μπορούν να, να συμμετέχουν σε δημοπρασίες, να μην μπορεί κανείς να εκφράσει επιθυμία, να συνεχίσει ή να συμμετάσχει σε δημοπρασίες, γιατί η μαφία προβαίνει σε δολοφονίες και έτσι καταλήγουμε τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται αντικείμενο κατάχρησης. Πολλά χρήματα από τα γεωρικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταλήγουν τελικά να αξιοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για τις υποθέσεις αυτές και ίσως η Κομισιόν μπορεί να μας ενημερώσει περαιτέρω για αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι και ο Όλαφ έχει ήδη αναλάβει δράσεις. Θέλουμε να μάθουμε και ποια βήματα έχει κάνει η Κομισιόν. Η Κατερίνα έχει έρθει σε επαφές με την οικονομική αστυνομία της Ιταλίας, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και καθόλου, μα καθόλου εύκολη. Το αντίθετο, είναι επικίνδυνη η δουλειά αυτή να δώσω το λόγο στην κυρία Μπόρχμαν που είναι και η αγαπημένη μας σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση. Παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Έχω και καινούριο μικρόφωνο. Συγγνώμη, εξεπλάγει λίγο γιατί νόμιζα ότι θα δίνατε το λόγο πρώτα στον, στον Όλαφ γιατί μιλάμε για πάτη. Αν θέλετε, ναι, παρακαλώ, ας δώσουμε το λόγο στον ε, Όλαφ πρώτο. Είμαστε απόλυτα ευέλικτοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Όποιο ε, θέλει τον λόγο πρώτο, α τοποθετηθεί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χριστίνα, ευχαριστώ που μου παραχώρησε τη σειρά σου. Όσον αφορά τα γεγονότα για τα οποία έχουμε διαβάσει όλοι στα ΜΜΕ, αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι μια υπόθεση την οποία διερευνούμε ως Όλαφ. Αποτελεί όμως τμήμα μιας ευρύτερης ανησυχίας, αν θέλετε, ε, μιας σωρίας ε, εκθέσεων και αναφορών και υποθέσεων που παρακολουθούμε. Όπως γνωρίζετε, ο Όλαφ δραστηριοποιείται και έχει αναλάβει δράση σε πολλές υποθέσεις στο παρελθόν, σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές, με την Οικονομική Αστυνομία της ε, Ιταλίας και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Οικονομική Αστυνομία της Ιταλίας ε, υπάρχουν βεβαίως και οι καραμπινιέροι και οι εισαγγελικές αρχές που κάνουν εξαιρετική δουλειά για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων. Θα θυμάστε βεβαίως ότι έχουμε ως Όλαφ συντάξει εκθέσεις σχετικά με όμοιες, παρόμοιες υποθέσεις στο παρελθόν και θα ήθελα να σας ε, αναφέρω τι θεωρούμε ως σχεδόν φυσική εξέλιξη στην απάτη σε αυτό τον τομέα οι γεωργικές πληρωμές, όπως και κάθε ε, κονδύλια που δίνονται ε, αποτελεί πηγή έλξης ε, για απάτης και σε αυτή την περίπτωση εγκληματιών. Εδώ βεβαίως ακόμη περισσότερο γιατί είναι χρήματα χωρίς ε, κίνδυνο. Αυτά θέλουν οι εγκληματίες. Χρήματα χωρίς μάλιστα να διατρέχουν και κανέναν κίνδυνο. Βλέπουμε στην πορεία του χρόνου πως ε, φαινόμενα που σχετίζονται με τον εκφοβισμό ή ακόμη και την άσκηση βίας γίνονται αντικείμενο αναφορών πλέον και αυτό συνδέεται κατά τη γνώμη μας με το γεγονός ότι οι ενωσιακές ενισχύσεις σήμερα συνδέονται με την ιδιοκτησία της γης που δεν είναι ε, αφ' κάτι κακό γιατί στο παρελθόν είχαμε πολλές περιπτώσεις όπου οι πληρωμές συνδέονταν με την παραγωγή τη γεωργική. Κάτι που ήταν ακόμα χειρότερο όσον αφορά την προσέλκυση απάτης. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αυτό προφανώς θέλετε και σήμερα να συζητήσουμε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα προστατεύσουμε τον ενωσιακό προπολογισμό εναντί αυτών των περιπτώσεων απάτης και εναντί αυτών των εγκληματιών. Τα σημάδια που παίρνουμε ε, είναι ενθαρρυντικά δεν χαιρόμαστε βεβαίω που υπάρχει η απάτη, όμως είναι υγιές το γεγονός ότι γίνεται έρευνα. Διότι αυτό σημαίνει ότι εντοπίστηκε η απάτη αυτή από τις ιταλικέ αρχές και ότι ε, αναλαμβάνονται βήματα για την καταπολέμησή της. Κάτι που μας χαροποιεί. Σημαίνει ότι με, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το σύστημα λειτουργεί. Αν βεβαίως θα είναι η τελευταία υπόθεση σχετική που θα μας απασχολήσει, η απάντηση είναι μάλλον όχι. Πρόκειται για μια συνεχή, έναν συνεχή αγώνα. Οι εγκληματίες, ξέρετε, είναι πολύ δημιουργικοί άνθρωποι και πολύ γρήγορα και εύκολα ξέρουν να εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Για να εξασφαλίσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ως σύστημα και για να άξιος να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν αδυναμίες γνωστές που δεν ε, εντοπίζονται και δεν αντιμετωπίζονται. Έχουμε βεβαίως ε, στενή συνεργασία και με την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας, θα σας τα πει και η Κριστίνα, αλλά έχουμε συνεργασία και με την Ιταλική αστυνομία και με τη δικαστική εξουσία της ε, Ιταλίας για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει συνεχής ανταλλαγή όλων των πληροφοριών που έρχονται στα χέρια μας. Υπάρχει λοιπόν ένας δια, διάλογος και μια ροή πληροφοριών που οδηγεί και σε καλά αποτελέσματα όπως αυτό που συζητούμε σήμερα. Να σταματήσω εδώ για να δω αν υπάρχουν ενδεχομένως και ερωτήσεις που θα θέλατε να μας απευθύνετε και που αφορούν όλες τις υποθέσεις που έχουμε διερευνήσει. Θέλω κλείνοντας απλώς να πω ε, να σας επιστήσω την προσοχή σε μια παλιά υπόθεση στην έκθεση 17, ε, την υπόθεση ε, Μπονίφικα, έκθεση του Όλεφ, που δεν ήταν ακριβώς η ίδια, απλά είναι χαρακτηριστική για το πώς εξελίσσεται η απάτη στην ε, πορεία του χρόνου. Πλέον, από τις πιο κλασικές περιπτώσεις εικονικών γεωργών, δηλαδή ενισχύσεων που ζητούνται για εκτάσεις γης που βρίσκονταν μέσα σε αεροδρόμια ή από νεκρούς. Όλα αυτά έχουν βελτιωθεί, δεν τα βλέπουμε πια τόσο. Ε, χάρη και στη δουλειά της, ε, του Όλαφ και της δουλειάς που έχουν κάνει οι συνάδελφοι από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και των σχετικών συστάσεων. Αλλά φαίνεται ότι πλέον μετακινούμαστε από την απάτη που αφορούσε την έκταση, η οποία, την ενίσχυση για μια έκταση που ζητούσε κάποιος νεκρός ή που βρισκόταν μέσα σε αεροδρόμιο, πλέον κινούμαστε σε, μια, σε, ένα νέο φαινόμενο πιο κλασικού εκφοβισμού από την πλευρά της ε, μαφίας, που επίσης είναι ένα ε, ε, φαινόμενο που πρέπει να καταπολεμηθεί στεναρά και βεβαίως ε, μόλις ξεκινήσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δουλειά της θα είμαστε ε, ένας από τους εταίρους που θα συνεργαστούμε συνολικά για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόρχμαν και στη συνέχεια η κυρία Κινίτσι έχει ζητήσει το λόγο. Thank you, Chair, and thank you for... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο μετά την Όλαφ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τις Ιταλικές αρχές και ιδίω την Guardia di Finanza, την, ε, την ε, οικονομική αστυνομία της Ιταλίας. Ε, και πέραν της περίπτωσης, δεν μπορώ να σας πω ότι έχουμε και πολλές πληροφορίες, γιατί είναι μια ποινική έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη στην Ιταλία και η πρώτη φυσικά που θα ενημερωθούν είναι η Όλαφ. Και εμείς όμως παρακολουθούμε την πρόοδο και προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε ότι όντως θα ανακτήσουμε τα χρήματα για οποιαδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, όπως είπε και ο συνάδελφος από την Όλαφ, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ δεν πρόκειται απαραίτητο για μια υπόθεση στην οποία αυτοί οι οποίοι απέκτησαν τη γη με τρόπο που δεν θα έπρεπε ε, παραβίασαν κανόνες της ΚΑΠ, όπως για παράδειγμα τα, ο άρθρο που είχαμε ε, στο Πολίτικο σήμερα το πρωί που λέγεται ότι κατά πάσα πιθανότητα η, η γη είναι ακαλλιέργητη και οι δορυφορικές φωτογραφίες θα μας πούνε αν όντω υπάρχει συντήρηση της γης και αγρανάπαυση ή όχι. Το θέμα είναι αν είναι επιλέξιμη η γη, σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται έχει αγοραστεί η γη με απαράδεκτο τρόπο αν θέλετε και είναι πιο δύσκολο να πούμε ότι είχαμε παραβίαση κανόνων της ΚΑΠ, αλλά σίγουρα έχει υπάρξει παραβίαση κανόνων. Και εδώ θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ποινική δίωξης στην Ιταλία. Όσον αφορά τώρα προηγούμενες υποθέσεις, περιπτώσεις στις οποίες αναφέρθηκε και ο κύριος Μπιάνκι. Υπήρχαν και θέματα που αφορούν ε, τον Ιταλικό Οργανισμό Πληρωμών, την ΑΤΖΕΑ, που είναι και ο οργανισμός ο αρμόδιος για την Ιταλία και εκεί ελήφθησαν συγκεκριμένα μέτρα. Η αρμόδια αρχή στην Ιταλία έθεσε σε ε, ε, αναστολή τον οργανισμό πληρωμών και απομακρύνθηκαν άτομα τα οποία θεωρήθηκε ότι δεν είναι έμπιστα και αξιόπιστα μετά από την έρευνα της Όλαφ και μετά ε, υπήρχε ένα νέο σύνολο κανόνων ε, που συστήθηκε για τον οργανισμό πληρωμών. Τα παρακολουθεί αυτά η Γενική Διεύθυνση Άγκρη και καταγράφησαν πάρα πολλά χρέη μετά από αυτή την υπόθεση Μπονίφικα και ε, η Γενική Διεύθυνση Άγκρη κάνει δημοσιονομικέ διορθώσει, ώστε όλα τα χρήματα να επιστραφούν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Αν δείτε τι δημοσιονομικέ διορθώσει την τελευταία δύο-τρία χρόνια θα δείτε ότι έγιναν πάρα πολλέ διορθώσει για την Ιταλία. Στην ουσία είναι παλιά χρέη τα οποία σχετίζονται με κάποιε περιπτώσει ε, ε, που διαπιστώθηκαν στο παρελθόν, απάτη και έγιναν δημοσιονομικές διορθώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι δεν έχουν ανακτηθεί τα χρέη και δεν έχουν καταγραφεί καταλήλω στο Ιταλικό σύστημα. Οι Ιταλικέ αρχέ τώρα έχουν εξετάσει όλα αυτά τα χρέη και όλε τι υποθέσει και την υπόθεση Μπονίφικα, αλλά και σε συνεργασία με τη Guardia di Finanza ήταν ποια θα έπρεπε να είναι τα ποσά ε, τα οποία θα έπρεπε να ανακτηθούν και έγιναν δημοσιονομικέ διορθώσει για την Ιταλία. Για την υπόθεση τώρα που είναι σε εξέλιξη και αναφέρθηκε στο πολίτικο σήμερα, θα πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών των Ιταλικών αρχών. Θα ήθελα επίσης ε, να τονίσω και πάλι ότι δεν είναι βέβαια καλό παράδειγμα, αλλά είναι πάντα καλό να διαπιστώνει κανείς ότι οι εθνικές αρχές λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να παρακολουθούν τέτοιες απάτες και πλέον ε, εξετάζουν το θέμα και εμείς θα παρακολουθούμε και τυχόν πρόοδο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις. Κατερίνα πρώτα. Και μετά θα συνεχίσουμε. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους εκπροσώπους της Όλαφ και της Κομισιόν για αυτά τα οποία μας είπανε αλλά βεβαίως ε, και για την εκτίμηση που εξέφρασαν για τις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας μου, οι οποίες ε, αποκάλυψαν μια σοβαρή περίπτωση απάτης στο θέμα της χρηματοδότησης Γεωργίας. Η επιχείρηση ε, αυτή διεξήχθη στην Σικελία, ονομάστηκε Νέμπροντι. Ε, σε συνεργασία με την εισαγγελία κατά της μαφίας και της τρομοκρατίας και εκεί πέρα οι καραμπινιέροι μαζί με την Guardia di Finanza έκαναν πολλές ε, συλλήψεις ε, και έκλεισαν επιχειρήσεις και δεσμεύθησαν επίσης πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ ε, που ήταν όπως είπαμε το ποσό της ε, απάτης. Όλα αυτά λοιπόν είναι αποτέλεσμα έντονων προσπαθειών ε, των διοκτικών αρχών, συγκεκριμένα της οικονομικής αστυνομίας, που έχει τις σχετικές αρμοδιότητες ε, της ε, δικαστικής αστυνομίας οπωσδήποτε τον αρμοδίο για την καταπολέμηση του ξεπλήματος ε, χρήματος και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μαφιόζικο οργανωμένο έγκλημα το οποίο έχει αναγνωρίσει και η Europol υπάρχει στην Ευρώπη και ε, στην χώρα μας και στην ε, Σικελία. Πρόκειται λοιπόν για ένα έγκλημα το οποίο χαρακτηρίζεται και σωστά υπόθηκε από τους εκπροσώπους της Όλαφ και της Κομισιόν από μια όλο και μεγαλύτερη επέκταση στον τομέα της ε, οικονομίας και θα ήθελα να αφαιρθώ και σε μια προσωπική μου ιστορία γιατί όπως ξέρετε ήμουν δικαστής, ε, κόρη δικαστή που δολοφονήθηκε από την μαφία το 1983 τον Ιούλιο ακριβώς γιατί είχε αντιληφθεί την βαρύτητα της ε, μαφιόζικης δραστηριότητας και το ότι ε, μπαίνει πλέον και σε άλλους τομείς και προκαλεί ε, τεράστιες ζημιές. Λοιπόν, ακριβώς ε, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι έκφραση αυτής της τάσης του οργανωμένου εγκλήματος να εισέρχεται δηλαδή ε, να πηγαίνει εκεί όπου υπάρχουν τα λεφτά και μετά προχωράει σε ξέπλυμα του χρήματος, σε επανεπενδύσεις για να χρηματοδοτήσει και άλλες εγκληματικές ε, δραστηριότητες. Τούτου λεχθέντος λοιπόν θεωρώ πως η χώρα μου επέδειξε ακόμη φορά την ε, δυνατότητα να αποκαλύπτει τις απάτες προκειμένου τις οικονομικές να νομοθετεί σωστά, να έχει τα αντισώματα θα έλεγα γιατί όπως σας είπα από την περίπτωση του πατέρα μου έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια και έχουν αναπτυχθεί τα αντισώματα ή η κατάλληλη νομοθεσία, μια δικαιοσύνη η οποία έχει τεταμένη την προσοχή της, η αστυνομία η οποία παρακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές, οπότε έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, να αποκαλύψει τις απάτες, αυτό είναι το βασικό, και να τις αντιμετωπίσει επαρκώς και πράγματι ε, θα περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα της ε, έρευνας, αλλά ήδη νομίζω πως ε, τα αποτελέσματα είναι ήδη σημαντικά. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στα λόγια του εισαγγελέα το Καφιεροντέρα ο οποίος ήταν ε, παρόν σε μία εκδήλωση και ήθελε να τονίσει το πως σε όλα τα κράτη-μέλη ή το οργανωμένο έγκλημα με την διαφθορά, με τη μαφιόζικη μέθοδο του εκφοβισμού, των απειλών, της βίας και της ε, διαφθοράς, με το ξέπλυμα του χρήματος, με τις απάτες, τις ευρωπαϊκές πληρωμές ε, εις χωρίς το οικονομικό σύστημα εις βάρος των ε, συμφερόντων της κοινότητας βλάπτοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό την επιχειρηματικότητα και το ερώτημα είναι ακριβώς ε, ποιος ε, θα μπορέσει να αντιταχθεί σε αυτό το οποίο απομακρύνει και τις υγιείς ε, επιχειρήσεις. Ακριβώς λοιπόν έλεγε ο εισαγγελέα ότι πρέπει να εξεχρονίσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα ήθελα ακριβώς να επαναλάβω τα λόγια του, τα οποία τα είπε ξεκάθαρα νομίζω, γι' αυτό θα ήθελα να τα επαναλάβω. Τόνισε ότι εάν δεν δράσουμε αποφασιστικά για να αντιταχθούμε στο οργανωμένο έγκλημα, στην μαφία, θα τους ε, επιτρέψουμε να ε, μπορέσουν να ελέγξουν την ε, οικονομία. Θα πρέπει ακριβώς άρα σε όλα τα επίπεδα να αντιταχθούμε στο οργανωμένο έγκλημα το οποίο παρεμβαίνει στην οικονομία και στα δημόσια οικονομικά των χωρών μας και της Ένωσης. Μία σκέψη ακόμα. Έχουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2017, την έκθεση την σχετική ε, αναγνώρισε λοιπόν εκεί πέρα πως η Ιταλία είναι μεταξύ των κρατών μελών ε, τα οποία είναι πιο δραστήρια όσον αφορά την ανείχνευση ε, και την καταγγελία τέτοιων περιστατικών στην κοινή γεωργική πολιτική. Και η Κομισιόν καλεί να συνεχίσουν να στηρίζονται τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί και ο αριθμός και η ποιότητα των ελέγχων και να ανταλλαχθούν οι βέλτισες πρακτικές ε, στον τομέα αυτό και νομίζω ότι η Ιταλία μπορεί να διαδώσει τις βέλτισες πρακτικές εδώ πέρα γιατί η επιχείρηση αυτή η οποία αποκάλυψε αυτές τις απάτες είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, μιας εμπειρίας ε, συσσωρευμένης ε, και αυτό οφείλεται δυστυχώς στο ότι αντιμετωπίζουμε το οργανωμένο έγκλημα στην πιο βίαιη μορφή του στη δεκαετία 70 και 80 και ποτέ δεν έχουμε χαλαρώσει και προσπαθούμε ακριβώς στον τομέα τον νομοθετικό και τον δικαστικό να βρούμε τους τρόπους ε, για να πολεμήσουμε την μαφία η οποία συνεχώς ε, εισχωρεί στον τομέα αυτό πρέπει και στο ευρωπαϊκό επίπεδο να ενταθεί το σύστημα των ελέγχων οπωσδήποτε και προληπτικά Ήδη η εκπρόσωπος Κομισιόν ανέφερε κάποιες από τις σχετικές ε, πρωτοβουλίες ε, και οπωσδήποτε να αρχίσει να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εγκαίρως ε, και να έχει τους απαραίτητους πόρους πρέπει να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή των πληροφοριών να ενισχυθεί η ανταλλαγή των οικονομικών πληροφοριών, να ανταλλαχθούν οι βέλτιστες πρακτικές και να περάσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιταχθούμε στη μαφία, την ευρωμαφία όπως ήδη ε, υπόθηκε. Θα σταματήσω εδώ, θα ήθελα όμως ε, να επαναλάβω αυτό το οποίο είπε και η κυρία Χολμάερ. Θα ήθελα να προτείνω στην Επιτροπή μας ε, να κάνουμε μία αποστολή στην Ιταλία για να δούμε απευθείας την κατάσταση της χώρας, να συναντήσουμε τους ανθρώπους εκεί πέρα, την εισαγγελία κατά της μαφίας και της τρομοκρατίας, την οικονομική αστυνομία που είναι εξειδικευμένοι σε αυτά τα ζητήματα και για να εντείνουμε τις σχέσεις μας ε, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η χώρα μου λοιπόν έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν καταστάσεις ε, δραματικές αλλά συνεχίζει τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Οπότε είναι καλοδεχούμενη η στήριξη της ε, Ένωσης ε, και ακριβώς ε, η στήριξη από την Επιτροπή μας σε όλα τα επίπεδα για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απάτες οι οποίες δεν ξέρω αν περιορίζονται μόνο σε έναν κλάδο, ας πούμε, αν η ΚΑΠ τους ε, ελκύει ιδιαίτερες. Ε, επισέρχονται παντού και πάρα πολύ συχνά εκεί όπου υπάρχουν ε, χρηματοδοτήσεις. Οπότε θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα. Σας ευχαριστώ. και επαναλαμβάνω την πρόσκλησή μου για να έρθετε στην Ιταλία και να έρθετε σε άμεση επαφή με τους ε, οργανισμούς ε, επιβολής ε, του νόμου σε όλους τους κλάδους και όσον αφορά βεβαίω και τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Καταρίνα. Ήσουν πολύ καλά προετοιμασμένη. Έχω ορισμένες ερωτήσεις με τον γενικότερο τίτλο που αποτελεί και μια δήλωση του επικεφαλής της Ιταλικής Αστυνομίας λέει ότι έχουν βρει νέους δρόμους για την εξασφάλιση πλούτου που βάζουν στην τσέπη τους χωρίς να υπάρχει κίνδυνος. Και ενώ συντηρούν κλασικές ε, οδούς ε, αποκόμισης ε, πλούτου όπως είναι τα ναρκωτικά και τα όπλα έχουν ε, ένα και περισσότερο αξιοποιήσει και την απάτη κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα λέω αυτά διότι δεν μας απασχολούν μόνο ζητήματα όπως αυτά που μας απασχόλησαν στην στη Σλοβακία και στην Ιταλία, αλλά μιλούμε πλέον και για θέματα ιδιοκτησίας. Πρόκειται για εκτάσεις που ανήκαν στο κράτος. Δεύτερον, οι δημοπρασίες που έγιναν έγιναν αντικείμενο απάτης με τον εξής τρόπο. Με το που εμφανίζονταν ονόματα γνωστών οικογενειών της μαφίας, δεν τολμούσε κανείς άλλο να συμμετάσχει ή να υποβάλει προσφορά, γιατί προφανώς κανείς δεν θέλει να δολοφονηθεί, να φάει μια σφαίρα στο κεφάλι γιατί έκανε ε, τη λάθος κίνηση σε δημοπρασία. Οπότε το, το ερώτημα είναι γιατί δεν μπαίνει μέτρα, στο κράτος, μέτρα το κράτος να έχουν ενδεχομένως μια ε, ιδιαίτερη μεταχείριση οι, οι, αγρότες που έχουν γειτονικά αγροτεμάχια. Ε, γιατί είναι πρόβλημα να μην μπορεί κανείς να συμμετάσχει σε μια δημοπρασία επειδή φοβάται ότι θα, θα δολοφονηθεί. Οπότε πρόκειται για μια μορφή προσετερισμού ε, ιδιοκτησίας με τον οποίο, τον οποίο δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης τα κέρδη από αυτές τις δραστηριότητες είναι τεράστια ακριβώς γιατί η αγορά ήταν, ε, η, η τιμή αγοράς ήταν ελάχιστη η, και η συνολική τα συνολικά έξοδα λειτουργίας ε, ενός τέτοιου αγροτεμαχίου είναι πάρα πολύ ε, χαμηλά. Πώς μπορεί κανείς να το επιτύχει αυτός, με, αυτό, με, με δουλειά, με μαύρη εργασία προσφύγων. Πώς ακριβώς καλλιεργείται τελικά η γη αυτή. Γιατί ε, βλέπουμε ότι τυπικά όλοι οι κανόνες της ε, ΚΑΠ τηρούνται. Με ενδιαφέρει αυτό. Πώς μπορούν τα, να είναι τόσο υψηλές τα, κέρδη από τις ε, ενισχύσεις ε, βάσει της έκτασης, γιατί έγινε πάρα πολύ δουλειά για να καθοριστούν τα κριτήρια με τα οποία μπορεί κανείς να λάβει ενίσχυση ένας κανονικός ε, ε, γεωργός χρειάζεται να ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις, ε, σε αυτά τα κριτήρια, σε αυτές τις προϋποθέσεις. Από ό,τι φαίνεται το οργανωμένο έγκλημα δεν δεσμεύεται από αντίστοιχες υποχρεώσεις, καταφέρνει και τις ξεπερνάει. Πώς ακριβώς γίνεται. Βλέπω και στη Σλοβακία και στην Ιταλία ότι όλο ένα και περισσότερο ο παράγοντας που καθορίζει το πώς διαμορφώνονται τα πράγματα είναι η πίεση που ασκείται παρασκηνιακά και στην Τσεχία είχαμε αντίστοιχε υποθέσει. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει κατά κύριο λόγο να συζητήσουμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε ή πρέπει να πάρουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα φαινόμενα. Είναι κλασικές ε, μέθοδοι ε, Εξαπάτηση του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε άλλους τομεί. Στη Γεωργία είναι σχετικά ε, ε, πρωτοφανέ να χρησιμοποιούνται αυτές οι μέθοδοι. Βλέπω ότι γίνονται τέτοιες έρευνες και σε άλλους τομείς. Υπήρξε και η σκέψη, η σκέψη να κάνουμε ένα, μια αποστολή στην Καλαβρία και στη Σικελία γιατί για άλλη μια φορά ο τοπικός πληθυσμός πλήττεται από τέτοια φαινόμενα. Και πρέπει νομίζω και να δώσουμε κι εμείς ένα πολύ στεναρό μήνυμα για την αντιμετώπιση. Θα το συζητήσουμε στους ε, ε, συντονιστές βέβαια πρωτού πάρθει μια απόφαση. Ο κύριο Αστέλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Όλαφ και τη Γενική Διευθυνσία Άγκρη για τα στοιχεία τα οποία μα έδωσαν. Ε, παρά το γεγονό ότι αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή υπάρχει ποινική έρευνα σε εξέλιξη δεν μπορούμε να έχουμε ε, τα ακριβή στοιχεία αυτή τη ιστορία. Να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Κινίτσι. Όλα όσα μας είπατε μας βρίσκουν σύμφωνους, ε, ε, ειλικρινά. Ε, συμφωνώ επίσης κυρία Πρόεδρε και με τις δικές σας τις γενικές παρατηρήσεις, ε, διότι θα πρέπει να μας απασχολούν και αυτά πέραν των όσων ανακάλυψε ο Ιταλός εισαγγελέα, ε, το, ε, το γεγονός ότι αυτές οι πρακτικές φαίνεται να είναι πολύ πιο συχνές από ό,τι ε, μας δίνεται να καταλάβουμε. Είναι συχνές γιατί είναι απλές, είναι και χονδροειδείς ε, ως προς πρακτικές, αλλά είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές ε, και φυσικά επικερδείς και αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί. Θα πρέπει να ανησυχεί σε δύο πτυχές. Καταρχάς, ο Ιταλός εισαγγελέα και οι Ιταλοί ανακριτές ε, θα πρέπει τελικά να ε, πατάξουν μια πρακτική ε, που αποσυντονίζει ουσιαστικά εσωτερικά τη χώρα. Τελικά από όλε αυτές τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις Πώς καταλήγουμε όλες αυτές οι πρακτικές της μαφίας να περνάν από όλο το σύνολο των ελέγχων που έχουν ήδη ε, χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την επαλήθευση των τίτλων ιδιοκτησίας. Πραγματικά εκπλήσωμαι που διαπιστώνω ότι μια τέτοια οργάνωση σε τέτοια κλίμακα ε, δεν μπόρεσε να διακρίνει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι ακόμα σε λειτουργία. Και φαίνεται ότι η έλεγχη που έχουμε δεν αρκεί. Και θα έπρεπε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί ει βάθο, προκειμένου να έχουμε πολύ πιο αποτελεσματικά συστήματα. Και η δεύτερη πτυχή είναι μια πτυχή υποθετικής διάστασης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μια τόσο απλή και επικερδής ε, πρακτική και μια πρακτική η οποία τελικά δεν ε, ε, προϋποθέτει και πολλές, ε, πολλούς κινδύνους για αυτούς που τη χρησιμοποιούν. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί η χρήση αυτής της πρακτικής σε όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και διασταυρούμενοι έλεγχοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις ενισχύσεις ε, που δίνονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ε, και που λαμβάνουν ε, για γεωργικές εκμεταλλεύσεις, διότι μπορεί να ανακαλύψουμε και πολλά επί του ζητήματος. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια σκέψη για την ε, δημιουργία μαύρης λίστας σε δημοπρασίες για εκτάσεις γης. Γιατί αν είναι σαφές και γνωστό ότι σε μια περιοχή δραστηριοποιούνται ε, οικογένειες της ε, μαφίας, τότε πραγματικά ε, πώς γίνεται να επιτρέπουμε αυτές οι οικογένειες να λαμβάνουν μέρος σε τέτοιες ε, δημοπρασίες, να μην αποκλείονται δηλαδή όταν έχει αποδειχθεί ότι γίνεται κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε μάλλον το θέμα της ιδιοκτησίας και το ποιος τελικά καλλιεργεί τις εκτάσεις αυτές. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ναι, επειδή ε, πολλά από τα ερωτήματα ε, αφορούσαν το τι κάνει η Κομισιόν και τι μπορεί να γίνει. Θα υπενθυμίσω αυτό που είπε ο συνάδελφος Μπιάνκι. Μπορούμε να πούμε ότι οι πρακτικές έχουν εξελιχθεί. Έχουμε ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο δεν, παλιότερα δεν λειτουργούσε πολύ καλά στην Ιταλία, όσον αφορά αυτούς τους εικονικούς γεωργούς, αλλά και εκτάσεις που δεν ήταν επιλέξιμες. Εκεί έγιναν βελτιώσεις στο σύστημα ε, ελέγχου. Ξέρετε, μέσω δορυφόρου μπορούμε να διαπιστώσουμε πολύ εύκολα ποιε εκτάσεις είναι ε, επιλέξιμες και ποιε όχι. Έχουμε ε, χαμηλές, χαμηλά σφάλματα σε, την, σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει όμως η, η, μετά η εξή κατάσταση. Υπάρχει ε, επιλέξιμη έκταση, αλλά το θέμα είναι πώς έχει κανείς καταλήξει να είναι ιδιοκτήτης, κάτοχος αυτής της έκτασης ως ενοικιαστής, ως ιδιοκτήτης. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα ελέγχου μας λειτουργούν πολύ σωστά για να διαπιστώσουμε αν καλλιεργήθηκε μια έκταση. Όταν λέει το άρθρο στο ε, πολίτικο ότι δεν υπήρχε πολύ κίνδυνος, ε, χρειάστηκε ωστόσο να καλλιεργηθεί αυτή η γη, όχι να υπάρξει συγκεκριμένη παραγωγή η ενίσχυση ε, αναεκτάριο στην Ιταλία κατά μέσο όρο είναι 3,27. Κάποιες φορές οι αρχές πληρώνουν περισσότερο γιατί αν υπάρχουν, αν υπάρχουν οπορώνες για παράδειγμα τότε τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αλλά πρέπει κανείς να καλλιεργήσει τη γη. Δεν μπορεί να πας να φυτέψεις δέντρα και να σηκωθεί να φύγεις. Πρέπει να διατηρείς την ε, πρόεδρος διακόπτη. Ναι, εγώ έθεσα ε, ε, ερώτημα για τη δουλεία που είναι γνωστό φαινόμενο στην περιοχή. Ναι, απαντά η εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Με βάση του κανόνε επιλεξιμότητα ε, τη ΚΑΠ, η γη καλλιεργήθηκε. Πώ καλλιεργήθηκε και από πού προήλθε το εργατικό δυναμικό και πώ ε, περιήλθε στην, περιουσ... στην ε, κατοχή αυτών που... των οποίων περιήλθε η, η γη αυτή, αυτό είναι ένα πιο περίπλοκο θέμα. Όταν κανείς υποβάλει αξίωση ε, στην Ιταλία ε, για ενίσχυση, πρέπει να αποδείξεις ότι ε, σου ανήκει η γη ή ότι την νοικιάζεις νόμιμα. Και κοιτάζουμε εμείς με τους δορυφόρους μας αν πράγματι διατηρείται η γη αυτή. Τώρα, αν το κάνουν δούλοι αυτό, τότε δυστυχώς στην ΚΑΠ δεν έχουμε πλέον κανόνες για να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Αυτό αφορά τους εθνικούς κανόνες που καταρτίζονται υπάρχει αυτή η διάκριση. διάκριση. Ε, εξαρτάται από το ποια είναι η νομοθεσία που παραβιάζει κανείς και φυσικά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει μεταφορά της ιδιοκτησ... του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ε, σε... με ρυθμό υψηλότερο από ό,τι ε, ήθιστε. Ε, εδώ πρέπει να δούμε και ζητήματα κατανομής της, ε, της γης. Εδώ δεν, δεν μπορούμε απλά να πούμε σε έναν οργανισμό πληρωμής «Κοιτάξτε το, αυτό το θέμα». Πρέπει συνολικά να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το νέο είδος παράκαμψης ε, που παρατηρούμε ε, όσον αφορά την απόκτηση ε, γεωργικών εκτάσεων. Βεβαίως, θα πρέπει κανείς να διατηρεί την γη. Ο κίνδυνος για το πώς θα αποκτηθεί αυτή η υγεία, η γη είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν ξέρω πώς θα απαντηθεί αυτό νομικά, γιατί μόλις κάποιος πει ε, ότι δεν μπορείς να κάνεις το ένα ή το άλλο πράγμα, υπάρχει κάποιος άλλος που θα καταφέρει να παρακάμψει αυτόν τον, ε, τον κανόνα. Δυστυχώς τον κανόνα δεν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή από πλευρά μου τουλάχιστον κάποια εύκολη λύση την οποία να μπορούσα να σας ε, προτείνω. Πάντως ε, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να το δούμε, να το βλέπουμε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και κάποιες προτάσεις που έχουν γίνει από την Καμισιόν ε, και στο πλαίσιο τη πρόταση για το ΠΔΠ, στον, στην κατηγορία τη στήριξη του κράτου δικαίου. Ίσως και αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να κρατήσουμε στο νου μας για το μέλλον. Και θέλω να πω και στην κυρία Κινίτση ότι την ευχαριστώ για όλες αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε για το τι γίνεται στην Ιταλία. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό παράδειγμα Περίπτωση όπου οι εθνικές αρχές ανέλαβαν δράση, αξιοποίησαν και την εθνική νομοθεσία προκειμένου να αντιμετωπίσουν ένα υπαρκτό, υπαρκτό πρόβλημα. Πρόεδρος, μου φαίνεται λίγο ότι η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε, δυστυχώς. Γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε τόσο τέλειοι και αποτελεσματική. Αλλά τι να κάνουμε, δυστυχώς ε, την, ε, την, ε, τη χώρα την έχει καταλάβει η μαφία. Τι να πω, προσπαθώ να το αντιμετωπίσω και εγώ με χιούμορ αυτό το θέμα. Το ζήτημα της, της δουλείας, της εργασίας υπό καθεστώς δουλείας είναι είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο της ΚΑΠ να μην υπάρχει κανόνα, κανόνας νομικού χαρακτήρα που να αποκλεί και να αποτρέπει τη χρήση δούλων ε, στις ε, εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και μάλιστα από εγκληματίες. Ίσως λοιπόν η Κομισιόν θα μπορούσε να σκεφτεί ότι ναι, παράγονται κάποια φρούτα αλλά ε, αν είναι να πεθαίνουν άνθρωποι για να καλλιεργούμε εμεί αυτά τα φρούτα, ε, κάτι πρέπει να μα προβληματίσει. Δεν λέω ότι αυτό κάνετε, ότι κλείνετε τα μάτια σα και δεν σα ενδιαφέρει το θέμα, αλλά δεν μπορεί να μα αφήνει αδιάφορου παγερά το θέμα ή τέλο πάντων καταγγελίες ότι άνθρωποι πεθαίνουν στις ε, καλλιεργήσιμες εκτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι διαφορετικά αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σκλαβιά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επιτύχει κανείς τόσο υψηλή κερδοφορία όπω αυτή που αναφέρεται στο πολιτικό. Και δεύτερον, η διοκτησία και ε, ε, ενοικίαση γης είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οπότε και εκεί θα, με, θα με ενδιέφερε αν ε, πρόκειται να αλλάξουν οι κανόνες στην Καλαβρία και στη Σικελία για το σε ποιον τελικά καταλήγει η χρήση της γης. Διότι αν οι οικογένειες είναι τόσο οικογένειες, οι οικογένειες είναι τόσο γνωστές, ώστε κανείς να μην τολμάει καν να, να, να προσπαθήσει να νοικιάσει μια συγκεκριμένη έκταση επειδή ξέρει ότι αυτή, αυτή την έκταση τη θέλει η μαφία ε, τότε ή οι, ε, οι τοπικές αρχές δεν είναι καλά ενημερωμένες ή υπάρχει ένα ευρύτερο σύστημα. Το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ένα τέτοιο φαινόμενο να εμφανίζεται. Έτσι όπως το περιγράφει και ο αρχηγός της αστυνομίας. Μα κάποιος πρέπει να ξέρει τι γίνεται. Δεν μπορεί όλοι να μην γνωρίζουν. Εμείς πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να μάθουμε. Υπάρχει εμπλοκή και κρατικών αξιωματούχων σε αυτό το κύκλωμα, σε αυτό το φαινόμενο. Ε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και από άποψη θεσμική και δομική στην Καλαβρία και αντιστοίχως και ο αγώνας για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων είναι δύσκολος, όμως πρέπει να γνωρίζουμε σε πρώτη φάση τι συμβαίνει ώστε να μπορέσουν οι αρχές, οι αστυνομικές, οι εισαγγελικέ αρχές να αντιμετωπίσουν και να ξεριζώσουν αυτό το θέμα. Ίσως θα μπορούσαμε να σκεφτούμε περισσότερα εργαλεία τα οποία θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας. Ίσως και όλα αυτά μπορούσαν να μας δώσει κάποιες σκέψεις. Πάντως σε κάθε περίπτωση εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά το θέμα, ώστε στην πορεία του χρόνου, καθώς θα συλλέγουμε και περισσότερες γνώσεις και πληροφορίες, να ξέρουμε και να μπορούμε να καθορίσουμε ποιε θα πρέπει να είναι οι επιπτώσεις όταν ανακύπτουν τέτοια ζητήματα κατοχής της γης, ενοικίασης ε, καλλιεργήσιμων εκτός, εκτάσεων και καλλιέργειας των ε, εκτάσεων. Και τι κάνουμε όταν εντός μιας χώρας δεν αρκούν από ό,τι φαίνεται οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί και τελικά μέσω δουλείας καταφέρνουν ορισμένοι εγκληματίε να επιτυγχάνουν τόσο υψηλά κέρδη. Διότι σε αυτόν τον κλάδο τέτοια ποσά δεν μπορεί κανείς να κερδίσει χωρίς δούλους, χωρίς σκλάβους, δεν μπορεί κανένας μικρομεσαίος αγρότης να επιτύχει τέτοια ποσά αν δεν χρησιμοποιούνται και τέτοιες δόλειες και παράνομες μέθοδοι όπως είναι η χρήση εργατικού δυνομικού υποκαθεστώς δουλείας. Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα να συνεχίσω ακριβώς από εκεί που σταματήσατε κι εσείς. Το... Και αυτό είναι και το βασικό ερώτημα πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο και γιατί τα αφήσαμε να συμβεί. Και θα ήθελα να επιστρέψω στην έννοια που σας παρουσιάστηκε προηγουμένως, που είναι το γεγονός ότι εξελίσσονται αυτά τα ε, εγκλήματα. Και ο μόνος ε, πραγματικός τρόπος που βλέπω από τη δική μας την πείρα να τα αντιμετωπίσουμε είναι η γνώση. Και νομίζω ότι έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Κινίτσι. Η ανταλλαγή πληροφοριών και οι βέλτιστες πρακτικές είναι ένας πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπος να εξασφαλίσουμε ότι σε όλη την Ευρώπη όλες οι αρχές γνωρίζουν τι συμβαίνει ώστε να μπορούν να το εξετάζουν. Ο κύριος Αστέλ ε, πολύ σωστά λέει ότι ε, δεν είναι και πολύ προηγμένο ε, σύστημα απάτη. Συνήθως η απάτη δεν είναι υψηλή τεχνολογίας. Το τέλειο έγκλημα είναι χωρίς κίνδυνο, πολλά χρήματα, αλλά πολύ απλό. Και αυτό που έμαθα από τη δουλειά μου τόσα χρόνια είναι αυτό. Αν ε, ε, ήμουν εγκληματικό μυαλό, θα μπορούσα να είχα σκεφτεί το σχέδιο στα 16 μου, χωρί πολλέ γνώσει. Και ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ω σύστημα, ω Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι ο εγκληματία δραστηριοποιείται σε ένα πολύ ενιαίο, ελεύθερο, ανοιχτό χώρο. Υπάρχει δικαιοδοσία, υπάρχει τομέα αρμοδιότητα, υπάρχουν σύνορα, υπάρχουν διάφορε αρχέ οι οποίε παρεμβαίνουν ταυτόχρονα. Και αν δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για αυτές τις γνώσεις και αν δεν μπορέσουμε να έχουμε τα πάντα να λειτουργούν αποτελεσματικά προς τη σωστή κατεύθυνση και η σωστή κατεύθυνση είναι ότι οι ε, εγκληματίες δεν θα ε, πρέπει να βάζουν στην τσέπη τους ε, τα χρήματα του δημόσιου κορβανά, δεν θα τα καταφέρουμε. Και νομίζω ότι το είπατε πάρα πολύ σωστά κι εσείς. Τίθεται θέμα διαχείρισης γεών, ιδιοκτησίας γεών και δεν είναι αυτό που έλεγε η συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Αγκρή, ότι έχει, δεν έχει σχέση με τη λειτουργία της ΚΑΠ, διότι αν πάω εγώ και πω στη μητέρα μου τι κάνω κάθε μέρα, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι η ΚΑΠ λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και ότι οι κανόνες κτήσης γης είναι τελείως διαφορετικοί και λειτουργούν διαφορετικά. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε όλοι ώστε να υπάρξει αυτή η συνεννόηση και να μην ε, ε, ε, παραγνωρίσουμε το γεγονός και ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο υψηλά, είναι υψηλά προηγμένο Το θέμα είναι ότι αν υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση που ελέγχει τη γη, κανένα δεν θα πάει στη δημοπράτηση τη γη. Ε, η κυρία Κινίτσι πολύ σωστά αναφέρθηκε στον έλεγχο τη περιοχή ε, από αυτέ τι εγκληματικέ οργανώσει. Και το αναφέρει και το άρθρο του Πολίτικο. Υπάρχουν περιπτώσει στι οποίε είσαι και ο ιδιοκτήτη. Δεν είναι, ε, συμμετέχει σε μια δημοπρασία και έρχεται κάποιο, που χτυπάει το κουδούνι, λέει. Θα του πει κράτα εσύ τις γιατί εγώ τι θέλω τη ζωή μου, ευχαριστώ πολύ. Και νομίζω ότι τίθεται και τέτοιο θέμα. Και ω Ιταλός τώρα μιλώ, δεν εκπλήσωμαι. Τα έχω δει πάρα πολλές φορές αυτά στα νιάτα μου και μεγάλωσα εγώ με αυτά τα φαινόμενα. Και με αυτά τα φρικτά εγκλήματα τα οποία διαπράττονται, δικαστές και εισαγγελείς που τα ερευνούν σκοτώνονται. Και η ουσία εδώ είναι ότι θα πρέπει να τα έχουμε όλα μαζί, να λειτουργούν από κοινού, τα συστήματα ελέγχων ε, και οι δικλείδες ασφαλείας και νομίζω ότι αυτό ε, συνέβη, αλλά δεν αρκεί για να αντιμετωπίσουμε τέτοια εγκλήματα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το ιταλικό μοντέλο υπάρχουν αυτοί οι υπερδικαστές οι οποίοι μπορούν τελικά να συγκεντρώσουν όλες τις γνώσεις σε εθνικό πλέον επίπεδο και πραγματικά ελπίζω ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας θα μπορέσει να κάνει κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή μαφία και το ευρωπαϊκό έγκλημα, το οποίο ελοχεύει ο κίνδυνο να δούμε ε, στη σήμερον ημέρα. Υπάρχουν και άλλε ιδέε, πολύ ωραίε ιδέε που άκουσα, ναι, μαύρε λίστε, αλλά για να φτιάξει κάποιο μια μαύρη λίστα χρειάζεται πληροφορίε και πρέπει να ξέρει και πού να ψάξει. Όταν εμείς ε, ερευνούμε στην Όλαφ ε, υποθέσεις ε, επιδοτήσεων που να ψαξει οταν εμεί πάρα πολύ μικρές η κάθε μία ξεχωριστά, πολύ μικρά ποσά, ε, χρειάζεται πολλή δουλειά για να ψάξει κανείς και πρέπει να ξέρει και πού να ψάξει. Και έρχομαι και πάλι εδώ στην έννοια της γνώσης, ανταλλαγής πληροφοριών και των πρακτικών. Και νομίζω ότι αν πραγματικά πάτε επί τόπου στην Ιταλία, θα μάθετε πολλά για το τι ακριβώς συμβαίνει και θα μπορέσετε να τα συνδυάσετε και με άλλα στοιχεία. Αλλά από τη δική μα την πλευρά, από την πλευρά τη Όλαφ, επενδύουμε ενεργά ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι γνώσει που έχουμε και γνώσει που αποκομίζουμε από συνεργασία με δικαστέ, με αρχέ, με οργανισμούς πληρωμής, ε, με υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι όλα σε ένα σημείο μαζεμένα, ώστε να μπορέσουμε και εμεί εύκολα να τα μοιραστούμε ευρύτερα. Ξέρω ότι δεν είναι η πανάκια, αλλά σίγουρα είναι ο καλύτερο τρόπο που βλέπω εγώ, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε κατάλληλα εξοπλισμένοι για να δώσουμε τη μάχη και να προσπαθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, αυτό όμως ε, σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κάποιων αρχών. Αλλιώς ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητες να αντιδράσουν οι οργανισμοί πληρωμών. Γιατί κοιτάνε όντω αν καλλιεργείται το έδαφος κτλ. Αλλά ότι ο άλλο είναι μαφιόζο ε, ε, ε, δεν μπορούν να το ξέρουν. Καλό είναι λοιπόν να σκεφτούμε πώς θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε αυτές τις πληροφορίες για τις μαφιόζικες δομές και οικογένειες. Και πράγματι δεν έχουμε βρει ένα σύστημα σχετικό. Γιατί δεν είναι και πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι η πολλωστή φορά. Ε, βλέπουμε ανθρώπους από στρατόπεδα προσφύγων στην Ιταλία που εργάζονται υπό συνθήκες σκλαβιάς, δεν ξέρω τα ονόματά τους κτλ είναι πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και θα έχουμε οπωσδήποτε και αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη δουλειά που κάνατε. Η κυρία Βίντσι έχει μία ερώτηση. Ε, εγώ αυτά τα ξέρω μόνο από την ε, τηλεόραση ευτυχώς ε, και δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω ε, συμβουλές αλλά νομίζω το ελάχιστο θα ήταν η τήρηση της εθνικής εργατικής νομοθεσίας και ο έλεγχος και βεβαίως ε, το θέμα των εποχιακών ε, την εποχή της σοδιάς είναι πάντα ένα θέμα να πληρώνονται σωστά θα πρέπει να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία τώρα για τις δημοπρασίες εμείς ε, πάντα θέλουμε περισσότερη διαφάνεια, αλλά στην περίπτωση αυτή μάλλον ε, θα έβλαπτε τους αγρότες, ε, γιατί θα γίνει γνωστό ότι λαμβάνουν ενισχύσει και άρα και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή όταν κάποιος ζητά ενισχύσεις και υπάρχει διαφάνεια, εμφανίζεται κάποιος και του λέει «Ωραία, δώσ' μου τα λεφτά τώρα». Πρέπει να το δούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι βλαβερή η διαφάνεια γιατί οι εγκληματίε ενδιαφέρονται για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ενημερώνονται. Είναι ακριβώς αυτό το προφίλ που περιγράφηκε πριν. Παίρνω 327 ευρώ, πώς θα γίνει με σκλάβους ε, να μπορέσω να καλλιεργήσω την έκταση αυτή ώστε και πώς θα μπορέσω με την χαμηλότερη δυνατή τιμή να αποκτήσω αυτή τη γη για να μπορώ να παίρνω αυτά τα 327 ευρώ ως ενίσχυση και να βγάζω και χρήματα από την ε, παραγωγή. Είναι εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα φυσικά και είναι ε, προφανώς ε, εύλογη η προϋπόθεση για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας αλλά βεβαίως ε, βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση πρέπει να είναι συνολικά η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Γιατί χωρίς ε, αυτό δεν μπορούμε να, να προχωρήσουμε ούτε να λύσουμε αυτά, αυτού του είδους τα φαινόμενα. Στη Γερμανία είναι προϋπόθεση να τηρείται η εργατική νομοθεσία και μάλιστα πρέπει και να αποδεικνύεις ότι τηρείς την εργατική νομοθεσία γιατί αν δεν το κάνεις έχεις πρόβλημα και δεν παίρνει και ενισχύσεις. Γιατί από ό,τι φαίνεται, όπως είπα και νωρίτερα, η θεραπεία πέτυχε, ο, νεκρός, ο, ο ασθενής απέθανε. Γιατί φαίνεται ότι στην ε, Ιταλία τελικά όλοι οι κανόνες, ακόμη και η τήρησή τους, δεν επαρκούν για να αποφεύγεται η τέλεση αξιόπινων ε, πράξεων. Όπως και να έχει, θα, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ όλους για την ε, συζήτηση που είχαμε. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή, ε, γιατί όπως λέγαμε και χτες, ε, δεν μας ενδιαφέρει να δυσκολέψουμε τη ζωή των, του 98% των κανονικών γεωργών, αλλά θέλουμε να εντοπίσουμε αυτό το 2% εκείνων που προβαίνουν σε πράξεις απάτης. Ich darf mich also dann... Λοιπόν, να, ευχαριστήσω και τον κύριο Μπιάνκι για την παρουσία του εδώ σήμερα. Ολοκληρώσαμε τα θέματα της σας διάταξης. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου, 2.30 με 6.30, 20 Φεβρουαρίου το πρωί και στις 5 Μαρτίου. Στο μεσοδιάστημα θα έχουμε και την αποστολή μας στην ε, Τσεχία, η οποία θα διαρκέσει δύο μέρες και στο πλαίσιο της οποίας θα έχουμε διάφορες ενδιαφέρουσες συναντήσεις. Α, και σήμερα το απόγευμα θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σε συνεργασία με την Επιτροπή ΑΦΚΟ στην αίθουσα 3Ε2, όπου θα μας συνοδεύσει ο κύριος Άνταμ και θα μας ε, παρουσιάσει μια έκθεση γύρω από το θέμα των πολιτικών κομμάτων και της χρηματοδότησής τους. Εγώ μίλησα ε, με τον άνθρωπο αυτό και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Γι' αυτό και θα πρέπει το θέμα αυτό να, συζητήσει, να συζητηθεί ε, και κλεισμένων των θυρών είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτή η έκθεση και κατά την έννοια αυτή θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να παρευρεθείτε σε αυτή τη συνεδρία. Σας ευχαριστώ πολύ και τα λέμε σήμερα το απόγευμα.